Bueno, Λοιπόν, ας αρχίσουμε σιγά σιγά διότι έχουμε ένα σημαντικό προσκεκλημένο που έχει και άλλα σημαντικά ε, σήμερα. Έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε στην Επιτροπή μας το Πρόεδρο Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ε, ο ΙΕ που είναι ο κύριος Γιώχη Ρούκερ, πώς προφέρεστε, Ρούκερ. Ρούκερ το λένε. Δεν ξέρω, με τις προφορές έχω πρόβλημα, μην προσβάλλω κανένα προσκεκλημένο. Λοιπόν, ας έχει. Στη Γενέβη είχαμε συναντηθεί με τον κύριο Πρέσβη και τον προσκαλέσαμε να έρθει στην υποεπιτροπή μας όταν θα ε, περνούσε από τις Βρυξέλλες, διαδραματίζει ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό, όπως όλοι γνωρίζουμε, στα Ηνωμένα Έθνη. Διευθύνει ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, με πάρα πολλά στοιχεία που του επιτρέπουν να έχουν ευρύτατη και βασίτατη αντίληψη για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απανταχού της γης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρίκερ που απεδέχθη την ε, πρόσκλησή μας και θα μας επιτρέψει να αναλύσουμε μαζί του τη σημερινή θεώρηση και προοπτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς το βλέπει ο ίδιος από τη θέση που κατέχει στον ΟΗΕ. Δεν θέλω εγώ να μακρηγορήσω, του δίνω μέσα το λόγο και τον ευχαριστώ απολύτως. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Υποεπιτροπής, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για μένα που είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Ευχαριστώ την Υποεπιτροπή σας που με προσκάλεσε μετά από την καποφόρο συνάντηση με την αντιπροσωπεία σας. Είχε έρθει με την κυρία Βαλενσιάνο, με τον κύριο Κρτσίμπ στην Γενέβη στην συνάντησή μας τον μήνα Μάρτιο. Και επίσης συναντήθηκα και με την Φεντερίκα Μογκερίνη ε, τον μήνα Μάρτιο σε υψηλότατο επίπεδο. Νομίζω ότι και η δική σας επίσκεψη και η επίσκεψη της Αντιπροέδρου, υπά της εκπροσώπου, υπογραμμίζει την προσπάθειά μας να υπάρξει ένα σύστημα πολυμερές στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς εκπροσωπείτε το μεγαλύτερο δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβουλευτικό σώμα στον κόσμο. Και το επαναλαμβάνουμε αυτό συνεχώς. Η συνεργασία σας με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της συμμετοχής των αντιπροσωπιών μας στις ολομέλειές μας είναι κάτι που εκτιμάται δεόντως στην Γενέβη. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί εντάσσεται και η επίσκεψή μου σήμερα, στενότερη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πριν σας ενημερώσω για την πρόσφατη συνάντησή μας, την 29η από τότε που δημιουργηθήκαμε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Το 2006 δημιουργηθήκαμε ε, προωθώντας ε, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις ή οδήποτε τύπου. Και όπως και η Υποεπιτροπή και το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών ασχολείται με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, ανά το κόσμο, ιδιαίτερα ε, καταγγέλλοντας και σημειώνοντας τις συστηματικές παραβιάσεις και κάνοντας συστάσεις επ' αυτών. Όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πριν 10 χρόνια ήταν τμήμα των μεταρρυθμίσεων της χιλιετίας και θα πρέπει να ειδωθεί και στα πλαίσια των υπολείπων πυλώνων των Ηνωμένων Εθνών, του πυλώνα ειρήνης, ασφαλείας, με κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις το 2005 μεταξύ των οποίων και της ανάληψης ευθύνης προστασίας ε, μαζί και με τον πυλώνα ευημερίας, οικονομικής ανάπτυξης και τους στόχους της χιλιετίας μετά το 2005. Έτσι λοιπόν και ο πυλώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα οδήγησε στην δημιουργία της, του Συμβουλίου αυτού. Γνωρίζετε ότι έχουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία θα θέσω ε, σύντομα. Νομίζω ότι οι συζητήσεις δημιουργούν, θα έλεγα, ένα πλαίσιο και ρίχνουν φως σε παραβιάσεις οι οποίες σε άλλες περιπτώσεις θα παρέμεναν στο σκότος. Είναι ένα μοναδικό πλαίσιο για να ακούγονται και οι φωνές από τη βάση, από τα κάτω, σχετικά με τις συστηματικές παραβιάσεις. Νομίζω η τελευταία μας ολομέλεια απέδειξε ότι αυτό το οποίο σκεφτήκαμε και δημιουργηθήκαμε για να κάνουμε, ε, αυτό ισχύει πλέον. Τώρα για την 21η περίοδο συνεδρίας, την οποία τελειώσαμε πριν μια εβδομάδα, ένα από τα βασικά θέματα μετά και από αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Είχαμε ένα διαδραστικό ενισχυμένο διάλογο για τα δικαιώματα αυτά των μεταναστών, τη συμμετοχή των εκπροσώπων της ΥΠΑ της και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δείχνει την ανταπόκριση του Συμβουλίου στις παρούσες κρίσεις και ανησυχίες. Η μετανάστευση συζητήθηκε από πολλές πλευρές και τα ανθρώπινα δικαιώματα έδωσαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν πολλές χώρες ότι η κρίση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σφαιρικά βλέποντας και ποιες είναι οι βαθιές αιτίες αυτών των μεταναστευτικών κινήσεων. Βλέπουμε παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προκαλούνται σε περιόδους και περιοχές συγκρούσεων, κοινωνικής και οικονομικής ανασφάλειας και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μοιρασμένη ευθύνη όλων των χωρών και των χωρών προέλευσης και των χωρών διαμετακόμισης και των χωρών κατάληξης ε, νομίζω ότι όλες εμπλέκονται με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Το Συμβούλιο υιοθέτησε δύο ψηφίσματα, το ένα αφορά τους εγκινήσει μετανάστες, τις μεταναστευτικές ροές και δεύτερον ε, τους εφήβους και τα παιδιά που μεταναστεύουν. Μια νέα πρωτοβουλία την οποία ξεκινήσαμε αφορούσε την ε, κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκα στη Μιανμάρ ζητήθηκε από την ο εκπρόσωπο να δώσει στοιχεία ιδιαίτερα για αναγκαστική μετανάστευση και εκμετάλλευση των μειονοτήτων των θρησκευτικών. Η κατάσταση είναι περίπλοκη σε επίπεδο μειονοτήτων στο Μιαμάρ, δεν αφορούν μόνο μία μειονότητα. Η κατάσταση χειροτερεύει, όπως είπε και ο ειδικός εισηγητής στην έκθεσή της. Υπάρχουν πολύ σοβαρά αντίμετρα τα οποία ελήφθησαν και τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια και τα παρατήρησε και η ίδια εκπρόσωπος. Θα αναφερθώ σε αυτά, τα αντίπεινα εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών. Το ψήφισμα το οποίο προωθήθηκε με όφηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μιανμάρ έχει σαν στόχο να τεθεί σε συζήτηση στο Συμβούλιο το θέμα αυτό. Ακούσαμε και την έκθεση της υπάτης εκπροσώπου. Είπε ότι τα κράτη οφείλουν στα πλαίσια ε, του κράτους δικαίου σεβασμό στους πολίτες τους και κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων υπήρξαν πάρα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα και υπογραμμίστηκε η ευθύνη των κρατών. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων μήνων. Τον Απρίλιο κάναμε το ίδιο σχετικά με τον Μπόκο Χαράμ και καταλήξαμε σε μια, ένα συνενετικό ψήφισμα το οποίο ε, αναφέρεται επίσης στην ευθύνη του κράτους στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Λοιπόν, για την τρομοκρατία υπάρχουν εφρικτά εγκλήματα στο όνομα της τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Αυτό μας απασχόλησε, υπήρξε διαδραστικός διάλογος με τον ειδικό εισηγητή από για τα θύματα της τομοκρατίας, των Μπεν Έμερσον έγινε και ένα πάνελ για τις επιπτώσεις της τομοκρατίας στα ανθρώπινα δικαιώματα και ενημέρωση για τις δράσεις και ε, τις κινήσεις του Μπόκο Χαράμ από τον Απρίλιο μέχρι τώρα. Οι ομιλητές όχι μόνο καταδίκασαν τις επιθέσεις της ομάδας αυτής εις βάρος κυρίως γυναικών και κοριτσιών, αλλά ζήτησαν από τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών τους. Ακούσαμε 21 παρουσιάσεις από εντολοδόχους ε, εισηγητές για θέματα όπως συνοπτικές εξελέξεις, φιλετικές διακρίσεις, άκρα παινία και περιορισμός ελευθερίας έκφρασης. Ακούσαμε και 14 εκθέσεις εργασίας της περιοδικής αναθεώρησης μεταξύ των οποίων και τις εκθέσεις Ισπανίας και Σουηδίας. Αυτό μας οδηγεί στην ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της διαδικασίας. Γιατί το UPR είναι τόσο σημαντικό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις απότερες περιοχές του κόσμου. Δημιουργήθηκε αυτός ο νέος μηχανισμός με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο εφευρέθη πριν 10 χρόνια όταν ακριβώς ε, τέθηκε σε λειτουργία το Συμβούλιο, να υπάρχει αυτή η περιοδική έκθεση και όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών ανά 4,5 χρόνια να υφίστανται έναν βαθύτατο έλεγχο των επιδόσεών τους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πράγματι το UPR που είναι τώρα στην τελική φάση του δευτερού του κύκλου όχι μόνο ε, επέτρεψε σε όλες τις χώρες να δείξουν πόσο ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο ε, αποδίδουν θα έλεγα, αλλά μας δίδει και ε, μέτρο για τον προσδιορισμό των βημάτων πρόοδου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς να μετρήσουμε, πώς να υπολογίσουμε την πρόοδο στον τομέα των διαφόρων συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε τις συστάσεις του πρώτου UPR με τις συστάσεις για το δεύτερο UPR και βλέπουμε πού έχει υπάρξει πρόοδος και πού έχει υπάρξει παναχώρηση. Ένα παράδειγμα για να το κατανοήσετε αυτό, η περίπτωση των νήσων Φίτζη. Σύμφωνα με την έκθεση για το Φίτζη υπήρξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο κύκλο. Ε, πήρε δραστήρια το Φίτζη μέρος στην Γενέβη και ακριβώς ε, στα πλαίσια της, ε, παραβι... της εξέτασης αυτής κατήργησε και τη θανατική ποινή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα παράδειγμα και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το UPR είναι ότι οι συστάσεις οι οποίες γίνονται και εδώ είμαστε σαν τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες υπέστησαν το UPR με πάνω των 50 συστάσεων. Σημαντικό είναι να αναπτύξουμε σωστά μέσα για τον υπολογισμό της εφαρμογής του UPR και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί ακόμα πριν ξεκινήσει ο τρίτος κύκλος. Επανέρχομαι τώρα στο Συμβούλιο στην τελευταία μας συνάντηση υιοθετήσαμε 25 ψηφίσματα και μία δήλωση του Προέδρου. Υπήρξαν δύο νέες εντολές, δύο νέοι εντολοδόχοι, ένας νέος εμπειρογνώμων για τους πολίτες της Αφρικής που υποφέρουν από αλμπινισμό γιατί διατρέχουν όπως γνωρίζετε οι αλμπίνο στην Αφρική υψηλού κινδύνους. Επίσης ε, το θέμα της ψηφιακής ε, ε, τεχνολογίας και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και ορίσαμε ένα ειδικό εισηγητή από τη Μάλτα. Να υπογραμμίσω επίσης ότι τα περισσότερα από τα κείμενα υιοθετήθηκαν με συνένεση παρά τις δύσκολες διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι το οποίο Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε και στο μέλλον όσο περισσότερη συνένεση γίνεται. Νομίζω ότι η πόλωση και ο ανταγωνισμός εμποδίζει να γίνουν γρήγορα τα πράγματα. Απαιτείται βέβαια συνοχή, πνεύμα συνεργασίας και διαλόγου. Αυτό το ονομάζω το πνεύμα της Γενέβης. Νομίζω ότι αν υιοθετήσουμε το 75% των ψηφισμάτων μας με συνένεση έχουμε ένα καλό ποσοστό. Σχετικά τα θεματολογικά τώρα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή δικαιώματα γυναικών, φιλετικές διακρίσεις επί τη βάση ε, της διαφοράς άνδρα-γυναίκας κτλ. Ε, συζητήσαμε το θέμα του δικαιώματος στην εκπαίδευση για κάθε κορίτσι και γυναίκα και της οικιακής βίας βάρος των γυναικών υιοθετήσαμε ένα σημαντικό ψήφισμα για την επιτάχυνση της κατάρχησης όλων των μορφών βίασης βάρος των γυναικών. Υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για τη διακρίση εις βάρος των γυναικών και χρησιμοποιούμε προχωρημένη ορολογία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά για τις γυναίκες. Υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις, δεν υπήρξε πάντα συνένεση, και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στον διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και συνεχίσει να είναι φαντάζομαι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη και στον χώρο, στον κόσμο. Τώρα, ε, είδαμε τι πετύχαμε με το ψήφισμα για τον Νότιο Σουδάν. Ε, παρά τις δυσκολίες ε, το Συμβούλιο τα κατάφερε και υπήρξε τελικά ενωμένο το Συμβούλιο στα πλαίσια των διαφορών. Και υπήρξε η συνένεση η επιθυμητή. Έγινε δεκτό λοιπόν το ψήφισμα ζητώντας να υπάρξει και μια ερευνητική επιτροπή και ε, για το Νότιο Σουδάν. Η ύπατη των Ηνωμένων Εθνών αποφασίστηκε να κάνει μια έρευνα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν και να πιέσει την κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν να συμμετέχει στις προσπάθειες να δράσει υπέρ της συμφιλίωσης. Ζητήθηκε από την ύπατη αρμοστία να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των βημάτων που έγιναν από την κυβέρνηση του South Σουδάν, της Νότιου Σουδάν. Συστήσαμε επίσης να υπάρξουν και για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δράσεις όπως τεχνική βοήθεια και διορισμός αν χρειαστεί ενός ειδικού εισηγητή. Να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο το πώς λειτουργεί η τεχνική βοήθεια ε, στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Πάρα πολύ συχνά γίνεται μια συζήτηση στο Συμβούλιο όπου οι ειδικέ καταστάσεις αναχώρα αντιμετωπίζονται με βάση το άρθρο 4 ή σύμφωνα με το 10 όταν συζητάμε τα θέματα της τεχνικής συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες. Ένας από τους δείκτες που συζητήθηκαν στα πλαίσια αυτά είναι τα κριτήρια έτσι ώστε να δούμε αν θα χρησιμοποιήσουμε το 4 ή το 10. Ε, προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση για τη βελτίωση της κατάστασης στη χώρα. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση τότε η απάντηση είναι το 10, αλλά αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση τότε χρησιμοποιούμε το 4. Για τη Συρία. Υπήρξε επίσης ένα ψήφισμα το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη για την ανάληψη ευθυνών για να σταματήσουν οι στρατιωτικές συγκρούσεις σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλες τις πλευρές. Ξέρετε ότι η βάση δεδομένων την οποία δημιουργούμε για τη Συρία είναι πληρεστάτη και περιλαμβάνει και τα ονόματα των υποτιθέμενων δραστών, έτσι ώστε κάποια στιγμή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί συχνά είναι η βάση των συζητήσεων και σε άλλα βήματα όπως το Συμβούλιο ασφαλείας τα συμπεράσματα της Επιτροπής μας δηλαδή. Για την Ουκρανία επίσης έγινε λόγος, δυστυχώς η πρωτοβουλία αυτή όμως δεν έτυχε συνένεσης, αλλά πέρασε σε ψηφοφορία με πλειοψηφία και πρέπει να υποβληθεί προφορική πρόταση ή σύσταση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία και τώρα προβλέπεται τακτική ενημέρωση στο Συμβούλιο. Πρέπει επίσης να σας πω ότι άρχισε και μια άλλη μορφή των σχέσεων υπά της αρμοστίας με το Συμβούλιο εκτός από τις τακτικές συνεδριάσεις τετραμηνιές προσπαθήσαμε για πρώτη φορά να δημιουργήσουμε και μία άτυπη μορφή συνεννοήσεων στη Γενέβη στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή και έτσι νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη καλύτερη ανταπόκριση προς καταστάσεις απρόβλεπτες παραπάνω από ό,τι δηλαδή οι συζητήσεις στις τακτικές συνεδριάσεις ή τις έκτακτες. Για την Λευκορωσία το Συμβούλιο ανανέωσε την εντολή του ειδικού εισηγητή στη 32η Σύνοδο και στην 71η στην Λευκορωσία, για τη Λευκορωσία. Εκτός αυτού, όπως ξέρετε ή ίσως διαβάσατε, η Επιτροπή για την Γάζα δημοσίευσε την έκθεσή της. Είχε κάνει διαβουλεύσεις με πολλούς μάρτυρες και θύματα στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα. Και η έκθεσή της έλεγε ότι μπορεί να πρέπει να δημιουργηθεί μια επιτροπή για εγκλήματα πολέμου α, εκ μέρους και Ισραηλινών και Παλαιστινιακών ενόπλων ομάδων. Η, στην υπάτη αρμοστία εγκρίθηκε ψήφισμα για το θέμα που ζητούσε από τον ύπατο να κάνει δική του έκθεση στην 31η Σύνοδο της Υπάτης τον Μάρτιο του 2016. Η Επιτροπή Έρευνας για την Ερυθρέα παρουσίασε επίσης την εκτενή της έκθεση 500 περίπου σελίδων, μπορεί μερικοί να την έχετε δει, για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν σε απερίγραπτη έκταση που σπανίως έχουμε δει αλλού και ενέκρινε και ένα ψήφισμα που ζητάει την επέκταση της Επιτροπής Έρευνας με ειδική εντολή για να συλλεχθούν αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση και να μαθαίνει τι συμβαίνει η πάτη αρμοστία. Τώρα, σύντομα να μιλήσω για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Σας είχα πει και από την αρχή ότι η πάτη αρμοστία από τότε που ε, δημιούργησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πριν από 10 χρόνια περίπου είχε προτείνει την ε, καθολική περιοδική αναθεώρηση ή έρευνα ή έκθεση για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και αυτό δεν είναι κάτι διακοσμητικό για μας, είναι βασικό γιατί δεν μπορούμε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας εάν δεν έχουμε αν δεν έχουμε πληροφορίες για την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο στο Συμβούλιο, στο ΣΑΔ, αλλά και αλλού. Και πληροφορίες από περιφερειακές και τοπικές μήκη οργανώσεις και συστήνουμε βασικά πράγματα που θέλουμε να συνεχίσουν να θεωρούνται βασικά για να διασφαλιστεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και να σχετίζεται με τις εργασίες του Συμβουλίου. Είτε επιτόπου στις διάφορες χώρες, είτε όταν υπάρχει κάποια διάδραση με το συμβού, κόσμο με το Συμβούλιο επισκεπτών στη Γενέβη κλπ. Και εγώ ως πρόεδρος του, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να παρακολουθώ πολύ λεπτομερώς οποιαδήποτε περίπτωση και προσπαθούμε συνεχώς να δημιουργούμε κάποια συνένεση στο Συμβούλιο γιατί όλοι έχουμε την ίδια αντίληψη ότι η κοινωνία των πολιτών είναι κάτι ουσικό, βασικό για μας και θέλουμε να μην το θεωρήσουμε διακοσμητικό. Αυτή είναι βέβαια και η ευθύνη μας και η εντολή μας αλλά πολύ σημαντικό και για την Προεδρία μου δεν θέλουμε να μειωθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, αντίθετα να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί. Τώρα για το μέλλον, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τη σημασία των ψηφισμάτων μας πέραν της εθούσης 20 του, του, στο κτίριο της Γενέβης, θέλουμε να πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επιπτώσεις όλων αυτών που κάνουμε θα είναι εγγυημένες στην αρχή της προεδρίας μου προσπάθησα να ταυτίσω τρεις, τρία, τρεις προτεραιότητες που αφορούν το, τα θεσμικά. Πρώτον, να βελτιώσουμε περισσότερο τις σχέσεις του, των δύο τμήματων του ΟΗΕ στη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη αλλά να λύσουμε και το χρηματοδοτικό πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε ο πυλώνας ανθρωπίνων δικαιωμάτων παίρνει μόνο 3% του προϋπολογισμού του ΟΗΕ, το οποίο είναι κάτι πολύ λιγότερο από ότι οι άλλοι πυλώνες για την ευημερία ή για την ειρήνη κτλ. Ο ύπατος αρμοστής βέβαια είναι και αυτός εν γνώση όλων όσων λείπουν αλλά προσπάθησα και εγώ να ταυτίσω την αποτελεσματικότητα, ποια είναι η αποτελεσματικότητα του ΣΑΔ, διότι δεν πρέπει να γίνουμε θύματα της επιτυχίας μας. Οι πρωτοβουλίες μας, ψηφίσματα, συζητήσεις, ειδικοί εισηγητές, ε, αυξάνονται, οι δραστηριότητες αυξάνονται γεωμετρικά και πρέπει να κάνουμε κάτι για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, όχι κάθε αυτή η αποτελεσματικότητα για την αποτελεσματικότητα, αλλά για να είμαστε ακόμα πιο λειτουργικοί με περισσότερα αποτελέσματα. Έγινε κάποια πρόοδος στους πρώτους μήνες για τις σχέσεις Νέας Υόρκης Γενέβης, όχι αρκετή ακόμα. Επίσης εγκρίναμε μία προεδρική δήλωση για την αποτελεσματικότητα και στην 29η Σύνοδο και για τη δεύτερη εξαμηνία περίοδο της Προεδρίας νομίζω ότι θα τονίσουμε περισσότερο το θέμα αυτό της αποτελεσματικότητας επιτόπου. Ιδιαίτερα για τον τρίτο κύκλο. Maybe I'll leave it at that. Thank you very much. Ίσως να σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε για τις τελευταίες εξελίξεις και θα δούμε τη συνέχεια. Ναι, ναι, όχι, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ήταν εκτενέστατη, εξαντλητική η παρουσίασή σας. Και είμαι βεβαία ότι και οι συνάδελφοί θέλουν να σας κάνουν ερωτήσεις. Η κυρία Μπίλερ πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά για αλλαγή και πιο γρήγορα θα συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για την παρουσίασή σας, για το πώς εργάζεται το Συμβούλιο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνετε. Ασχολείστε με πάρα πολλά πράγματα. Αν τα δούμε εμείς από πλευρά μας, ε, αυτές οι ε, περιοδικές ε, επισκοπήσεις UPR είναι πάρα πολύ χρήσιμες και στο Κοινοβούλιο κάνουμε ψηφίσματα για διάφορες χώρες, π.χ. για τη Σαουδική Αραβία. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι πολύ συχνά κοιτάμε τι έχει δεχτεί η χώρα και πόσο έχει προχωρήσει σε σχέση με τα όσα λέγονται και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για μας και πάρα πολύ χρήσιμα. Τώρα, έχω συμπραγματικές ερωτήσεις, διευκρινιστικές. Περιγράψατε ποια ήταν τα ψηφίσματα της τελευταίας συνεδρίασης. Γνωρίζετε πώς έχει η κατάσταση στη Βυρμανία και για τους Ροχίνγκα. Το Κοινοβούλιο έχει πληθώρα ψηφισμάτων περάσει και θα το συνεχίσουμε. Εγώ δεν έχω τώρα μεγάλη πληροφόρηση για τα ε, δικαιώματα των Ρωμά παγκοσμίω και το σχετικό ψήφισμα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εσωτερικό τη δηλαδή. Μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε τίποτα για το ψήφισμα και επίση τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Είναι κάτι που θα μα φανεί χρήσιμο στη δουλειά μα. Το φθινόπωρο νομίζω θα κάνει, ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ακρόαση μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών, διότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόβλημα. Ξέρετε ότι το πιο θανατηφόρο και επικίνδυνο σύνορο στον κόσμο είναι η Μεσόγειος. Δεν είναι δυνατό αυτό. Μιλάμε για αξίες από τις οποίες εμφορούμεθα. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, μια τέτοια πολιτική. Θα πρέπει να αξίζει το όνομά της αυτή η πολιτική των σύνορων με ανθρωπιά. Βλέπω ότι στην ημερήσια διάταξη ε, θα σας απασχολήσει αυτό το θέμα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη συνεδρίαση. Θα ασχοληθείτε με την Καμπότζη και ένα ε, θέμα που έχει να κάνει με την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα. Και στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχει συζητηθεί ε, ο τρόπος των παραβιάσεων εκεί των ανθρωπινών δικαιωμάτων και τι είδους παραβιάσεις χαρακτηρίζεται αυτό ενδεχομένω και ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Θα δώσετε κάποια συνέχεια και τέλος, εμείς που είμαστε περιφερειακός οργανισμός, κοιτάμε τι γίνεται και σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Π.χ. τι κάνει η Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική. Ήδη έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην περιφερειακή του ολοκλήρωση. Αλλά στην Νοτιοανατολική ανατολικη Ασία, ΑΣΕΑΝ, δεν έχουμε ακόμα πάρα πολύ ισχυρού δεσμού. Τι γίνεται εκεί, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πώ συνεργάζεται σε περιφερειακή βάση με διάφορου οργανισμού. Και τελευταίο, για τη χρηματοδότηση. Τώρα θυμάμαι ότι πληρώνουμε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ εδώ και χρόνια χωρίς να αυξηθεί την υποεποτροπή, υπογραμματεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά για το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων νομίζω εμεί δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση συμμετοχή σε αυτή. Μπορείτε να μα πείτε τι χρειάζεται να υποστηριχθεί. Και τώρα, στο επόμενο εξάμεινο, φθινόπωρο χειμώνα, θα καταρτιστεί μια έκθεση ε, για τη σχέση Ηνωμένων Εθνών Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έκθεση πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η ομάδα των φιλελευθέρων, αν δεν απατώμε. Έχετε σχόλια τι θα θεωρούσατε σκόπιμο και χρήσιμο να μπει σε αυτή την έκθεση, θα μας βοηθούσε τα μάλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λοχμπίλε, ο κύριος Χένκελ. Σενιόρ Χένκελ. Hm. Γεια σας κύριε Ρίκε. Την περασμένη φορά που σας είδα, Εργαζόμουν ήδη για τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς και εσείς ήσασταν πολιτικός. Πώς γυρνάνε τα στέφανα. Τώρα είστε εσείς ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικός είμαι εγώ. Έχω ερωτήσεις κάπως πιο θεμελιώδεις και ουσιαστικές. Είμαι εδώ ένα χρόνο τώρα και κάπως έχω σοκαριστεί πρέπει να σας πω από διάφορα που συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας ε, υπό δύο έννοιες. Πρώτον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε και εσείς την ίδια εμπειρία. Πρώτον, όλο και περισσότερο βλέπουμε να αυξάνεται και να διευρύνεται η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι εννοώ. Εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχουν ορισμένοι ε, εδώ στην Ομίγυρη που ε, προβάλλουν τα, τις ιδεολογικές τους αιμονές ε, και αγαπημένα τους θέματα υπό το των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Π.χ. η συζήτηση για τις αμβλώσεις. Είναι μια συζήτηση βεβαίως θεμητή ή ε, θέματα περιβαλλοντικά επίσης. Είναι θεμητό να τα συζητούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι ανήκουν κατά ανάγκη στην κατηγορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να σας δώσω ένα άλλο πολύ δραματικό παράδειγμα. Ανακάλυψα στην έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το έτος 2013 ότι ορισμένοι κατάφεραν να βάλουν ένα αίτημα για να μπει στην έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που για μένα είναι σκάνδαλο. Τι δουλειά έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα και όμως μπήκε στο κοινοβούλιο. Σας ερωτώ, πρώτον συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία μου ότι όλο και διονγκώνονται, διευρύνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα προς τον ορισμό τους που σε τελική ανάλυση ε, είναι μια επίθεση κατά των αρχικών στόχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μια δεύτερη ερώτηση, κάτι που έχω παρατηρήσει εδώ και χρόνια τώρα. Σε 55 από 57 Ισλαμικά κράτη τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται με τον α ή β τρόπο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κορίτσια και τις γυναίκες. Και ρωτώ, εσείς από τη θέση σας ή δεν ξέρω κάποιος άλλος ασχολείστε με αυτό το θέμα από ό,τι φαίνεται είναι εγγενές ε, η ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός της Ισλαμικής πίστης. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ανήκω σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τα δικαιώματα είναι αδιέρετα και σε αυτό το οποίο ορισμένοι ονομάζουν διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι το αδιέρετο είναι κάτι το δεσμευτικό εξ αρχής από την πρώτη διακήρυξη. Και αυτό δεν ερμηνεύεται πάντα με ισότιμο τρόπο και δίκαιο. Χαίρομαι λοιπόν που η περίοδος αυτής συνέλευσης αφιερώθηκε στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Έφτασα λίγο αργά ζητώ συγγνώμη και δεν άκουσα την αρχή της παρουσίασής σας κύριε Ρόκερτ. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε σε αυτό. Αν ναι παρακαλώ μπορείτε να επανέλθετε πάνω στα θέματα τα οποία έγιναν και αντικείμενο ψηφίσματος όπως το δικαίωμα στην κατοικία και το δικαίωμα στη διατροφή. Σχετικά με το δικαίωμα στη διατροφή νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του δικαιώματος στην ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως επίσης συνδέεται και με το θέμα της μετανάστευσης. Είμαι εισηγήτρια του θέματος της μετανάστευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες του Νότου της Ευρώπης και γι' αυτό παρακολουθώ τις εργασίες σας γύρω από το θέμα αυτό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανησυχώ λίγον για την διαίρεση που γίνεται ανάμεσα στις χώρες προέλευσης και στις χώρες διαμετακόμισης και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το δύσκολο να προσδιοριστεί πια είτε στο νότο είτε στο βορρά δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα γύρω από αυτό. Ομολογώ ότι εγώ δεν είδα το ψήφισμά σας για τα δικαιώματα των μεταναστών σε διαμετακόμιση, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό θέμα και γι' αυτό ακριβώς τα κράτη αυτά, τα κράτη διαμετακόμισης είναι και αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κάποιες χώρες του Βορρά γίνονται όλο και περισσότερο χώρες διαμετακόμισης. Ανήκω επίσης σε αυτούς που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ε, για την κατάσταση των χωρών στο κέρας της Αφρικής, στο Σουδάν και στην Ερυθρέα. Αν διάβασα καλά τις πληροφορίες, ο ειδικό εισηγητής για την Ερυθρέα έχει υποστεί απειλές κατά τη διάρκεια και του ίδιου του Συμβουλίου. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν λίγο περισσότερο για τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα για την Ερυθρέα και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε γι' αυτό. Για το Σουδάν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι τμήμα των επομένων θεμάτων στα οποία θα πρέπει να εκφραστείτε και θα ήθελα και εδώ να με φωτίσετε. Ο κύριος Μπασίρ. να ζητήσω συγγνώμη γιατί και εγώ καθυστέρησα να έλθω εδώ. Κύριε Ρούκερτ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε μπροστά μας εδώ σήμερα, αμέσως μετά από τον τερματισμό της τακτικής συνεδρίασής σας. Θα ήθελα να θέσω το θέμα των ε, προσώπων χωρίς πατρίδα, των απάτριδων. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους απάτριδες. Πρώτον, η ύπατη αρμοστία το Νοέμβριο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του φαινομένου αυτού τα επόμενα 10 χρόνια. Είναι πολύ καλός ο στόχος αυτός, όμως είναι σαφώς ότι αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση από πλευρά των εθνικών εταίρων και από πλευρά των υπολείπων πολιεθνικών οργανώσεων, τότε ο στόχο αυτό παρά είναι αισιόδοξο για να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, τι συγκεκριμένες δράσεις θα μα συστήσετε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των απάτριδων από τρίτες χώρες. Και το θέμα αυτό θα τεθεί ξανά στην ημερήσια διάταξη των εργασιών σας. Δεύτερον, ένα άλλο θέμα για μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα τους Μπιχαρή. Ξέρετε ότι η κοινότητα αυτή προέρχεται από την Ινδία, ζει στον Μπαγκλαντές κάτω από απαράδεκτες συνθήκες για δεκαετίες. Επίσημα το καθεστώς τους ε, έχει πλέον αναγνωριστεί και έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη του Μπαγκλαντές. Όμως παραμένουν για τους Μπιχαροί πάρα πολλά προβλήματα. Η ύπατη αρμοστία μου είπε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλοί Μπιχαροί οι οποίοι ε, φεύγουν με βάρκες από ότι υπάρχουν ροχίνγκα που φεύγουν με βάρκες για να πάνε σε άλλες χώρες. Λοιπόν, απαιτούνται περαιτέρω νομικές ρυθμίσεις στο Μπαγκλαντές είναι θέμα εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ευχαριστώ κύριε Μπεσίρ. Η κυρία Βέμπερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την παρουσίασή σας. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι πολύ υπέρ του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και οι αμφιβολίες μου για την, το όργανο αυτό αφορούν το πώς δημιουργήθηκε και τη σύνθεσή του. Πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά έχω πολύ μεγάλα προβλήματα να δεχτώ ότι χώρες που είναι γνωστές για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν παρακάθονται στο Συμβούλιο αυτό παρακάθυνται και κρίνουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες. Και γι' αυτό το ερώτημά μου είναι ναι ή όχι. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον μηχανισμό. Εγώ το σκέφτομαι, με ένα μηχανισμό που να βρίσκει ποιες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο αυτό και ποιες όχι. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Αλλά πρέπει επίσης να προσθέσω ότι για αυτά που είπε ο συνάδελφος, εγώ κάποτε δίδασκα ανθρώπινα δικαιώματα σε πανεπιστήμια και εξηγούσα πάντα στους φοιτητά μου ότι είναι αδιέρετα τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό είναι και καθολικά είτε μας αρέσει είτε όχι. Πρέπει να τα δεχτούμε όχι μόνο τα πολιτικά δικαιώματα αλλά και τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά. Και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί το θέμα της έκτρωσης ας πούμε τουλάχιστον όταν αφορά την ζωή της μητέρας, τον κίνδυνο της ζωής της μητέρας αν είναι αποτέλεσμα βιασμού ή Πώς μπορεί όλα αυτά να μην θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα, να μην θεωρεί ότι αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή τη γυναικεία αξιοπρέπεια και ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε το λόγο να ζητήσετε και θα σας δοθεί. Ε, κυρία Άντερσον. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Καθυστέρησα και εγώ, έχασα τα πρώτα λεπτά. Σας ευχαριστώ ε, που ήρθατε. Ξέρετε, εγώ είμαι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη και σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις μας διαβάσαμε την έκθεσή σας της 24ης Ιουνίου για την κατάσταση στη Γάζα. Καλωσορίζω τη δουλειά που έχει γίνει και τα λοιπά για την έκθεση αυτή, για την έρευνα, αλλά κάπως απογοητεύτηκα πρέπει να σας πω. Ε, γιατί από 3.000, 3.500 μάλιστα που σκοτώθηκαν στη Γάζα και ε, θέλω να πω ευθύ εξ αρχή ότι εγώ ε, καταδικάζω όλες τις επιθέσεις όποιες και να είναι αυτές και από όπου και αν προέρχονται. Αλλά νομίζω ότι αυτή η τακτική των ίσων αποστάσεων δεν είναι σωστή. Ε, αναφέρεται ε, κάποια ε, σχέδια για το πώς επιτίθεται το Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές, αλλά προκαλεί θανάτους οικογενειών ολόκληρων. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο τρόπο για ε, τέτοιες επιθέσεις από πλευράς Πανεπιστημίου στο Ισραήλ. Δεν είναι αντίστοιχες οι επιθέσεις. Ανησύχησα λίγο για τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει η διεθνής κοινότητα. Ήλπιζα να είναι πιο αποτελεσματική και πιο αποφασιστική στη δράση της. Και, και εκείνοι που ε, καταπάτησαν το διεθνές δίκαιο και ενδεχομένως έχουν ε, ε, διαπράξει εγκλήματα πολέμου δεν ξέρω αν έχουν ε, την ε, αντίστοιχη αντιμετώπιση. Και υπάρχει ένα διεθνέ δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται αυτό το θεμάτων και υπήρξε και μια σχετική απόφαση. Σα λέω, έχω απογοητευτεί από την έκθεσή σα γιατί τηρεί ε, τι ίσε αποστάσει σα δύο πλευρέ. Το Μάρτιο του 2016 θα εκδώσετε νέα έκθεση ε, για την ε, υλοποίηση και θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πώς συντάσσετε, πώς καταρτίζετε αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Ε, θα ήθελα κι εγώ. Μαρκαρέτε Άουκεν, είμαι εδώ. Είμαι αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπε η αξιότιμη πρόεδρος της αντιπροσωπείας μας. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγημε από αυτές τις ίσες αποστάσεις. Πραγματικά η αναλογικότητα είναι τμήμα της δουλειά σας, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στο σωστό τους ε, πλαίσιο και διάσταση. Ε, σε σχέση με αυτό που είπατε για τις μήκη οργανώσεις, έχουμε όλο και περισσότερα ε, παραδείγματα που διεθνείς ΜΚΟ παρεμποδίζεται. Η Μπάρμπαρα Μπίλερ είπε τι έγινε χτε στην Καμπότζη. πέρασε ένα νόμος ε, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τη διεθνή του υποστήριξη. Τι θα γίνει λοιπόν στο μόνο δημοκρατικό κράτο στη Μέση Ανατολή που είναι το Ισραήλ. Τώρα ε, προωθούν ένα νόμο σχέδιο που θα περάσει από την Κνεσέτ, το οποίο επί σε οργανώσεις όπως το Pet το Breaking the Silence που είναι οι Ισραηλινές οργανώσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν εξωτερική υποστήριξη χρηματική που δεν είναι και τίποτα τρελά λεφτά. Θα καταγραφούν και θα στιγματιστούν ως ξένοι πράκτορες. Ε, που, ε, αυτό είναι περίπου ταύτιση με εγκληματίες. Ακόμα και μία πρόταση ήρθε από κυβερνητικό κόμμα στην Κνεσέτ που είπε ότι θα πρέπει να φοράνε και δική κονκάρδα για να τους αναγνωρίζουν αυτούς τους ξένους πράκτορες. Αυτό το έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν με κάτι αστέρια. Και μας σοκάρει που το ακούμε τώρα ξανά. Και εγώ ανησυχώ και στεναχωριάμαι γιατί εξακολουθώ να θεωρώ το ε, Ισραήλ δημοκρατικό κράτος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, στεναροί ε, στο Λόγω και στη διατύπωση είναι θέμα τιμής. Το ξέρω ότι συζητάμε πολύ συχνά στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά προφανώς εξάρουμε και την καλή σας δουλειά και όλα αυτά. Αλλά τι γίνεται με, με, το, με οργανώσεις όπως είναι Vet και ε, Breaking the Silence, πάστε τη σιωπή, όταν τους φημώνουν και τους επιχρεώνουν να πάσουν, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε σε πολύ δεινή κατάσταση πραγματικά. Και τι θα γίνει με τους φίλους μας ιδιαίτερα. Okay. Ευχαριστώ κυρία Πόστη. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά που είπε η συνάδελφος Βέμπερ για το δικαίωμα των γυ... τα δικαιώματα των γυναικών επί του ίδιου των, του σώματος. Βρισκόμαστε στο 2015 και νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπερασπίσουμε την ιδέα μιας σύγχρονης κοινωνίας, μοντέρνας κοινωνίας. Επίσης θέλω να μας πείτε τι φρονείτε για το ψήφισμα που ανέφερε η κυρία Λόχμπιλντερ για τους Ρώμα. Γίνεται λόγο συνέχεια για δύσκολες καταστάσεις, για εγκλήματα παγκοσμίω. Εσείς τι κάνετε ως προς την πρόληψη γιατί μιλήσατε για το 3% του προϋπολογισμού του ΟΗΕ που δίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Ανεπαρκές αν θέλει κανείς πράγματι να εμποδίσει τη διάπραξη τέτοιων σοβαρών εγκλημάτων είτε από κοινού ανθρώπους είτε από πολιτικούς. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε την πρόληψη στα πλαίσια του ΟΗΕ. Νομίζω δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Θα δώσουμε το λόγο στον πρέσβη, ο οποίος έχει μεγάλο κατάλογο για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ja, tack så mycket. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις ερωτήσεις σας. Θα μιλήσω την Αγγλική για την ερώτηση της Λόχμπιχλερ και για τις δικές σας ερωτήσεις για τους Ρωμά. Δεν είχαμε τον Ιούνιο ψήφισμα για τους Ρωμά, αλλά είχαμε μία συζήτηση με τους ειδικού εκπροσώπους, εισηγητές για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την παρουσίαση μιας πρόσφατης μελέτης για την κατάσταση των Ρωμά. Συζητήσαμε επίσης ε, το φαινόμενο αυτό εις βάρος των ε, Ρωμά. So we did discuss, we didn't address it in a... στα αγγλικά, αν μεταφραστεί κατά λέξη, λέγεται αντιτσιγκανισμός, το βάζουμε σε εισαγωγικά. Τώρα για την Καμπότζη. Πρόσφατα, στην 28η ε, ολομέλειά μας, ορίσαμε ένα ειδικό εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη. Για τη Βόρεια Κορέα. Νομίζω ότι είναι βιτρίνα του πώς τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν σωστά σε σχέση ε, με τη συνεργασία μας με το Συμβούλιο Ασφαλείας. Υπήρξε μια Επιτροπή Έρευνας για τη Βόρεια Κορέα με πολύ θλιβερά αποτελέσματα όπως γνωρίζετε περιγράφοντας τρομερές ανησυχίες και παραβιάσεις και το Συμβούλιο Ασφαλείας τα συζήτησε αφού τα ψηφίσαμε εμείς. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια φυσικά συνδέονται. Υπήρξε η δυνατότητα επίσης παραπομπής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κάτι το οποίο νομίζω δείχνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την έννοια της απόδοσης ευθυνών γιατί δεν αρκούμεθα εμείς να τεκμηριώνουμε τις παραβιάσεις, αλλά απαιτείται και έλεγχος των πιθανών ενόχων. Γι' αυτό λοιπόν στην περίπτωση της Βορείου Κορέας και στα πλαίσια των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεχίσει να εξετάζει το θέμα και εμείς έχουμε ένα εισηγητή η ύπατη αρμοστία άνοιξε μια υπηρεσία στη Σεούλ για να παρακολουθήσει από κοντά την κατάσταση. Πολλά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και για πρώτη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας ήρθε στην συνάντησή μας τον μήνα Μάρτιο και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Δεν μας έπεισε βέβαια ούτε εμένα ούτε άλλους, αλλά αυτό που είπε δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα για τη συνεργασία με άλλες περιφέρειες. Αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση. Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία κάνει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία είναι να πηγαίνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, να έρχεται εδώ στις Βρυξέλλες. Εγώ πήγα στον ΟΑΣΕ και τη συνεδρίαση του μηχανισμού τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πάω και στην Άντις και νομίζω ότι η συνεργασία με περιφερειακούς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα δείχνουν την ανάγκη που υπάρχει ε, να συμμετέχει στις προσπάθειές μας η κοινωνία των πολιτών. Και αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τώρα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη παρατήρηση σύσταση να κάνω, όμως νομίζω ότι η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε με συμπληρωματικό τρόπο εν περιπτώσει και όχι με ανταγωνιστικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να το εφαρμόσει όπως το προβλέπει και η χάρτα στο άρθρο 8. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών παραδέχεται την ανάγκη την οποία υπάρχει ε, για συνεργασία σε όλους τους τομείς και στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη ε, και στη συνάντηση κορυφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ερώτηση Φίνκελ είναι πάρα πολύ θα έλεγα χρήσιμη για να δούμε αν πράγματι υπάρχουν πολλαπλές μορφές ορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάρα πολλοί ομιλούν για την πολυδιάσπαση της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση είναι θεμητή. Θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι όχι μόνο από την δήλωση της Βιέννης του 1993 αλλά και επί της ουσίας έχει υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα πολιτικά δικαιώματα από τη μία και τα πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα από την άλλη. Δεν πρέπει να υπάρχει εδώ παρανόηση. Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε είναι κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα συζητηθεί, σαν παράδειγμα στο περιθώριο του Συμβουλίου έχουν τεθεί θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών. Το δικαίωμα στο παιχνίδι είναι κάτι το θεμικό. Κανένα δεν μπορεί να είναι κατά του δικαιώματος στο παιχνίδι. Αλλά αυτή η πολυδιαφοροποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάπου θα πρέπει να σταματά. Πάντως εγώ δεν έχω να δώσω μια απάντηση εδώ ακόμα. Πάντως θα πρέπει επίσης να συμφωνούμε ότι σε επίπεδο ε, ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων ε, δεν πρέπει να υπάρξουν διακρίσεις. Αναφερθήκατε επίσης στα Ισλαμικά κινήματα στις μουσουλμανικές χώρες και στα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι θα πρέπει με όλες τις χώρες μας και, χώρα, τις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών εμένουμε στην καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε βέβαια να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό να κρίνουν όλες τις χώρες ότι κάτι συνιστά παράβαση ή όχι. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να συζητούνται και να αποφασίζονται. Η βασική αρχή στην οποία συμφωνούμε με όλες τις χώρες, όχι μόνο από το 1993 αλλά και από τότε συνεχώς, είναι ότι η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αδιαμφισβήτητη. Και όταν λέμε ότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία αυτών των δικαιωμάτων δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν θεωρεί ότι ισχύει η καθολικότητα. Μπορεί να ερμηνεύουμε με διαφορετικό τρόπο, μπορεί να εφαρμόζουμε με διαφορετικό τρόπο, μπορεί να παραβιάζουμε σαφώς τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σεβόμεθα πάντα το καθολικό χαρακτήρα ε, και το αδιέρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας. Είναι μια πολιτική παρατήρηση, ένα πολιτικό πρόβλημα και έχει μεγάλη σημασία. Εάν σαν παράδειγμα τέθηκε επίσης ένα άλλο θέμα και γίνεται μια συζήτηση για μια ευαίσθητη ισορροπία στο Συμβούλιο ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε ελευθερία πίστης και από την άλλη αυτό που ονομάζουμε και υπάρχει και ψήφισμα γι' αυτό ε, ο αγώνας εναντίον της έλλειψης ανοχής από πλευράς ε, των θρησκειών. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές. Κάποιες ομάδες χωρών είναι ιδιαίτερα έντονες σε σχέση με την έλλειψη ανοχής αυτή, τη μυσαλλοδοξία. Ε, κάποιες άλλες χώρες ε, ανησυχούν ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά και όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν σε βάθος, ιδιαίτερα με τους εκπροσώπους των μουσουλμανικών χωρών αλλά όλοι πιστεύουμε στον καθολικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό έχει σημασία. Θα συμφωνήσω ότι απαιτείται να ενισχυθούν από τη μία τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα από την άλλη. Σχετικά με τη μετανάστευση, Νομίζω ότι θα πρέπει να μελετήσετε τα ψηφίσματά μας και τις προτάσεις του ειδικού εισηγητού μας, του Φανσουά Κλερπό, για την Ερυθρέα. Τι είδου απειλές και αν υπήρξε απειλή εις βάρος του εκπροσώπου. Πράγματι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε στο ξενοδοχείο του και το υπογραμμίζουμε αυτό. Το Σουδάν παραμένει στην ημερησία διάταξη, έχουμε ψηφίσει αρκετά ψηφίσματα και θα συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το Σουδάν και όχι μόνο με το Σουδάν αλλά και με το Νότιο Σουδάν. Σχετικά με τους απάτριδες. Είναι στην ημερησία διάταξη εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν ψηφίσματα και στην 26η Ολομέλεια Υπάρχουν επίσης και εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την παράνομη στέρηση της ιθαγένειας. Συνεργαζόμαστε με την ύπατη αρμοστία και ε, υπό την καθοδήγηση του Αντώνιο Γκουτιέρες υπήρξε ένα πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση του φαινομένου των, ανθρώπων αυτών. Σημείωσα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπασίρ για τους Μπιχαρί. Θα ελέγξω τι ακριβώς γίνεται με τους Μπιχαρί. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στο UPR της Μπαγκλαντές και στο UPR της Μιανμάρα, στις εκθέσεις δηλαδή. Ε, δεν διαφεύγουν της προσοχής του Συμβουλίου τέτοιες περιπτώσεις και είμαι βέβαιος ότι και το συγκεκριμένο θέμα θα ληφθεί υπόψη στις συστάσεις μας. Σχετικά τώρα με την σύσταση του Συμβουλίου τα 47 χώρες μέλη ή 47 χώρες μέλη και λέγεται και στο, στην ιδρυτική μας χάρτα ότι θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μέγιστο βαθμό. Κατά κάποιο τρόπο κάνουν μια δήλωση ανάληψης υποχρέωσης όταν εκλέγονται στη Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε ότι το 1 τρίτο των μελών ανανεούται σε αιτήσια βάση ε, το φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη από τη Γενική Συνέλευση. Αλλά είναι μια Γενική Συνέλευση όπως πάντα η Γενική Συνέλευση ψηφίζει και λαμβάνονται υπόψη πολιτικές, ε, πολιτικά κριτήρια. Πάντως υπάρχει αυτή η ανάληψη υποχρέωσης από πλευράς των κρατών μελών και οι χώρες οι οποίες το κάνουν αυτό όχι μόνο πρέπει να σέβονται αλλά υπάρχει επίσης και ένα τμήμα της κοινωνίας των πολιτών που ελέγχει τις επιδόσεις των χωρών μελών. Για την έκθεση για τη Λωρίδα της Γάζα. Να πω ότι δεν είναι δική μας, το CUI είναι ανεξάρτητη οργάνωση. Εμείς σημειώνουμε τις εκθέσεις τους, τις υποβάλλουμε στο Συμβούλιο αλλά το CUI είναι όπως είπα ανεξάρτητο. Και αυτό είναι καλό. Σημειώνω αυτά τα οποία είπατε βέβαια για το ότι η έκθεση αυτή είναι αρκετά ισορροπημένη ή όχι τόσο ισορροπημένη. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε εξετάζοντας την έκθεση αυτή πάντως είναι ότι η αξιολόγηση στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι η έκθεση αυτή είναι πιο ισορροπημένη από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό το είδαμε σε πάρα πολλές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά για την Επιτροπή Έρευνας. Νομίζω ότι περίπου τα είπα όλα. Α, για τις ΜΚΙΟ. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ενίσχυση της παρουσίας των ΜΚΙΟ, έτσι ώστε να, να έχουν πάντα το χώρο που τους ανήκει να καταπολεμούμε τα αντίπεινα, να παρακολουθούμε τις αντιδράσεις εις βάρος τους, να δημοσιοποιούμε παραβιάσεις αυτές, ε, είπαμε για την ε, Ερυθρέα. Σε άλλες περιπτώσεις παρακολουθούμε μεμονωμένες ε, καταστάσεις ξεχωριστά και εγώ μεταφέρω όλες τις δράσεις μου για τα αντίπεινα στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος έχει στη διάθεσή του μια έκθεση για τα αντίπεινα αυτά εις βάρος των πρασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ επίσης και για το έργο σας. Ο πρέσβης προεδρεύει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου προφανώς οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ευρία πλειοψηφία. Και είδαμε και τις υπηρεσίες του και το επιτελείο του και ένα από τα καθήκοντά τους είναι να εξασφαλίζουν μεγάλες συνενέσεις ευρύτατες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι καθόλου εύκολη η κατάσταση στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Υπάρχουν μεγάλες περιφέρειες στον κόσμο που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο και έχουν και μεγάλη εξουσία και έχουν διαφορετική αντίληψη από τη δική μας εδώ. Ε, πάντως εκεί θα πρέπει να εργάζονται πάντα στα πλαίσια αυτά και καταπληκτικό έργο κάνουν και τους ε, συγχαίρομαι και υπόσχομαι ότι θα ξανάρθουμε να σας επισκεφθούμε το Μάρτιο. Ευχαριστώ πολύ.

Bueno, seguimos Συνεχίζουμε. Ha sido muy Πολύ ενδιαφέρον ε, αυτό το σκέλος της συζήτησης με τον πρέσβη. Πάμε τώρα στο επόμενο και θα συζητήσουμε για την προστασία των σχολείων καθώς επίσης και των πανεπιστημίων από την χρήση στρατιωτικών όπλων ε, από τις επιθέσεις, τις συγκρούσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που έκανε η Παγκόσμια Συμμαχία για την προστασία της ε, ε, παιδείας και της εκπαίδευσης σε εμπόλεμες ψηράξεις. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Υφυπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας είναι ο κύριος Hans Μπραντσκάρ από τους μεγάλους εμπνευστές αυτής της πρωτοβουλίας. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, για μένα είναι μεγάλη ικανοποίηση και τιμή που έρχομαι σήμερα να σας μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα για την Νορβηγική κυβέρνηση, την προστασία των σχολείων σε ένοπλες σειράξεις. Το θέμα όπως ξέρετε είναι κατεπήγον οι επιθέσεις κατά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε τουλάχιστον 70 χώρες συνέβησαν από το 9 μέχρι το 13 και από τότε συνεχίστηκαν. Γι' αυτό 37 εκατομμύρια παιδιά δεν μπορούν πια να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Σε μερικές χώρες το να πηγαίνει κανείς στο σχολείο είναι κάτι επικίνδυνο για ένα παιδί. Τα σχολεία υποτίθεται ότι είναι μέρη ελπίδας και μάθησης και όχι φόβου. Γιατί ε, τα σχολεία μπορούν να δώσουν ικανότητες και δεξιότητες στα παιδιά, στους νέους για το μέλλον. Τα ασφαλή σχολεία σημαίνουν και επένδυση για ένα ασφαλέστερο μέλλον και πιο μεγαλύτερη ευημερία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μεγαλύτερε προσπάθειε για να στηρίξουμε το δικαίωμα στην παιδεία ακόμη και σε καταστάσει σειράξεων. Η αναγνώριση τη ζωτική σημασία τη παιδείας για πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σημαίνει ότι η Νορβηγία αυξάνει τη συμμετοχή της σε τέτοια προγράμματα. Δεν θα είχε νόημα όμως αυτό αν δεν υπήρχαν δεσμεύσει για την προστασία των σχολείων κατά στρατιωτικών και άλλων επιθέσεων. Γι' αυτόν τον λόγο επιλέξαμε να είμαστε στην πρωτοπορία της διεθνούς προσπάθειας για την προστασία των παιδών σε περίπτωση σειράξεων. Ο μεγάλος αριθμός επιθέσεων κατά και πανεπιστημίων δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Με την Αργεντινή η Νορβηγία πέρυσι ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθηθούν κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία σχολείων και πανεπιστημίων κατά στρατιωτικών επιθέσεων, ενόπλων επιθέσεων. Έγιναν διαβουλεύσεις και μετά γράφτηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές. Οι συμμετέχουσες οργανώσεις και ορισμένα κράτη έπαιξαν το ρόλο τους και η Συμμαχία Οργανώσεων της ε, Κοινωνίας των Πολιτών συμμετέσχε και αυτή η Νορβηγία και η Αργεντινή αποφάσισαν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Έτσι με τις διαβουλεύσεις, οι διαβουλεύσεις κατέληξαν στην δήλωση για τα ασφαλή σχολεία. Οι διαβουλεύσεις τελείωσαν τον Μάιο φέτος. Στα τέλη Μαΐου η Νορβηγία τότε οργάνωσε στο Όσλο μία διάσκεψη για τα ασφαλή σχολεία όπου εκπροσωπήθηκαν 60 χώρες και πολλές μήκη οργανώσεις. Σχεδόν 50 χώρες μέχρι σήμερα δέχτηκαν αυτή τη δήλωση. Η δήλωση ασφαλών σχολείων ΔΑΣ σκοπεύει στην προστασία των όπλων και ιδιαίτερα των παιδών σε περίπτωση σύραξης. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ένα πρακτικό εργαλείο για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί διεθνώς για την προστασία των αόπλων και ιδίως των παιδών, μαθητών, φοιτητών και καθηγητών, καθώς και δασκάλων. Η δήλωση και οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι όμως επίσημα νομικά εργαλεία, αλλά έχουν δημιουργήσει μεγάλη η ε, ανταπόκριση διεθνώς. Ε, ελπίζουμε να μειώσει έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις επί της παιδείας της σειράξης. Πιστεύω κυρία Πρόεδρε ότι θα έπρεπε να σας περιγράψω τη δήλωση σύντομα. Στην αρχή αναφέρεται στα προβλήματα που προκύπτουν από τις ένοπλες σειράξεις και τονίζει τα πολλαπλά ωφέλη που μπορεί να αποφέρει. Μετά αναματίζει πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν κράτη και πολίτες σε καταστάσεις ένοπλης σύραξης και τονίζει τη σημασία που έχει η δουλειά και του ΟΗΕ για το ίδιο θέμα. Γιατί υπάρχουν ψηφίσματα και του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτό το θέμα. Η δήλωση αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και τις υποχρεώσεις να πάψει πλέον η ασυλία των ενόχων. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επίταξη σχολείων και πανεπιστημίων σε περίπτωση σύραξης ούτε αυτές είναι νομικά δεσμευτικές αλλά βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές. Αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην παιδεία, τη σημασία της προστασίας των αμάχων και τη δημιουργία ασφαλών σχολείων. Επίσης, συμφωνούν τα εξής. Χρήση των κατευθυντήριων γραμμών σε εθνικό επίπεδο και εφαρμογή τους από νομοθετικά εθνικά πλαίσια. Χορήγηση βοήθειας σε θύματα και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης παιδείας και διεθνής βοήθεια, υποστήριξη του ΟΗΕ για αυτά τα θέματα και τέλος τακτικές συναντήσεις αναθεώρησης των πεπραγμένων στην Ορβηγία. Ήδη έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε τις κατευθυντήριες και με συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρήσεις και αποσαφηνίζοντας τι πρέπει να γίνεται με στρατιωτικά κτίρια στο νορβηγικό έδαφος που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς σε καιρούς ειρήνης, διπλή χρήση όπως λέμε. Είναι και αυτός ένας τρόπος εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών που είναι αρκετά ευέλικτες για να εφαρμόζονται με διαφορετικούς τρόπους και να καθιστούν έτσι την παιδεία ασφαλέστερη. Η δήλωση για τα ασφαλή σχολεία έχει γίνει δεκτή από 47 μέχρι τώρα κράτη και είναι ακόμη βελτιώσιμη. Τον Μάιο έγινε η δήλωση του Όσλο και μπορούν όσα κράτη το επιθυμούν να προσθεθούν. Θα ήθελα τέλος να δηλώσω ότι η δήλωση δεν είναι το τέλος μιας διαδικασίας αλλά η αρχή της με κοινό στόχο την προστασία των σχολείων και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης σε περίπτωση σύραξη. Πρέπει να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε τα δικαιώματα των παιδών στην παιδεία. ώστε να γίνουν οι παιδες σύμβολα ελπίδας και όχι και τα σχολεία και όχι φόβου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε και την κυρία Άννα Σάστρε, που είναι η ε, διευθύντρια στην οργάνωση Save the Children, σώστε τα παιδιά. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μας δίνει την ευκαιρία work να μοιραστούμε μαζί σας μερικές σκέψεις για το πώς χρησιμοποιούνται τα σχολεία και τα πανεπιστήμια Save the Children ε, λέγεται οργάνωσή μας, Σώστε τα παιδιά ε, Παγκοσμίω εργαζόμαστε σε 120 χώρες και το 2014 είχαμε 55 εκατομμύρια παιδιά στα προγράμματά μας. Θέλω να αφαιρθώ σε ένα σημαντικό ζήτημα λόγω της απειλής που συνιστά για την εκπαίδευση. Η στρατιωτική χρήση των σχολείων είναι ένα φαινόμενο ευρέως διαδεδομένο. Στις περισσότερες χώρες που είναι σε ένοπλη σύραξη, 26 χώρες ήταν αυτές την περασμένη δεκαετία. Οι κυβερνήσεις ε, και οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών αλλά και αντάρτες χρησιμοποιούν τα σχολεία για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα χρησιμοποιούν ως στρατόπεδα βάσεις ε, εφοδιασμού, εποθήκες πυρομαχικών και όπλων, κέντρα κράτησης και ανάκρισης, ε, παρατηρητήρια κτλ. Ως υποδομή στρατιωτική. Και δεν παίρνουν μόνο τα σχολεία, αλλά και τα νηπιαγωγεία και κέντρα ημέρας σε χώρες όπως είναι η Συρία, το Νότιο Σουδάν και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Παίρνουν τα σχολεία και τα κάνουν στρατιωτικές βάσεις. Ε, όχι μόνο οι κρατικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και αντάρτικες ε, ένοπλες ομάδες απειλούν την ζωή ε, μαθητών και δασκάλων και καθηγητών. Άλλες φορές ε, καταλαμβάνουν πριν στο σχολείο και δεν αφήνουν τα παιδιά να μπουν μέσα. Αλλά πολύ συχνά χρησιμοποιούν ένα τμήμα μόνο του σχολείου, ενώ το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί ω σχολείο. Καταλαμβάνουν ένα όροφο, την αυλή ή μία αίθουσα. Έτσι ε, ε, εκθέτουν τους μαθητές στις επιθέσεις αντιπάλων ενόπλων ομάδων ή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Η στρατιωτική χρήση ενός σχολείου ε, μπορεί να ε, θέτει σε κίνδυνο το άμαχο καθεστώς ενός σχολείου. Και επίσης ε, υπάρχει κίνδυνος αντιπίνων. Χρησιμοποιούν επίσης και τα παιδιά ως στρατιώτες. Τα στρατολογούν ή τα χρησιμοποιούν ως βοηθητικό προσωπικό και μάλιστα ε, όχι μόνο παιδιά και γυναίκες ε, που υφίστανται και σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική βία. Εκτός από την ε, ασφάλεια των παιδιών υπάρχουν και καταστροφές στην υλικοτεχνική υποδομή και μακροπρόθεσμα μπορεί να επηρεάσει αυτό την εκπαίδευση γενιών ολόκληρων όπως βλέπουμε την εγκατάλειψη των σχολείων και ε, την ε, απομάκρυνση από την παιδεία για μεγάλες περιόδους. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε έκθεση για τους στόχους της χιλιετίας ε, το 2015 από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στις χώρες με ένοπλη σύραξη αυξάνεται από 30% το 99 που ήταν στο 36% το 2012 το ποσοστό των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο. Με το να πηγαίνει σχολείο μπορεί να σου σώσει τη ζωή. Το σχολείο μπορεί να αντιμετωπίσει τη ψυχολογική βία που ασκεί ο πόλεμο, να δώσει δεξιότητες και μόρφωση στα παιδιά και να τα προστατεύει από τη διακίνησή του στο τράφικινγκ από ένοπλες ομάδε. Ε, και μακροπρόθεσμα μια καλή εκπαίδευση σημαίνει ειρήνη και συμφιλίωση μετά τον πόλεμο και βοηθάει τα παιδιά και τους νέους να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται για να ε, φτιάξουν τη ζωή τους και την ευημερία στις ε, κοινότητες που ζουν. και δίνεται έτσι μια αίσθηση κανονικότητας, ομαλότητας ε, ε, στη ζωή τους ε, απέναντι στον πόλεμο. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τη δράση του Επιτρόπου Στυλιανίδη στην πρόσφατη σύνοδο κορυφή στο Όσλο για την παιδεία που είπε ότι η επίγουσα βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατευθυνθεί στην παιδεία. Υπάρχει ανάγκη για γραμμές για την προστασία σχολείων και πανεπιστημίων από τη στρατιωτική χρήση σε ε, καιρούς πολέμου είναι σημαντικό. Η Save the Children ε, μαζί με άλλους ε, εταίρους που έχουμε από όλο τον κλάδο έχουμε κάνει μια συμμαχία για να προστατεύουμε τα σχολεία από τις επιθέσεις και μεγάλη χαρά ακούσαμε την προθυμία της νορβηγικής κυβέρνησης να ηγηθεί σε αυτήν την προσπάθεια. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια συζητήσεων για να φτάσουμε εκεί ε, σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, διαφόρους κρατικούς και μη φορείς, ε, για να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να υλοποιηθούν. Και ε, οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν ακόμα, εκείνοι που κάνουν το στρατιωτικό σχεδιασμό ή έχουν επιφορτιστεί με τη διοίκηση για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα και τους κινδύνους. Επίσης, οι Υπουργοί Παιδείας και οι Υπουργοί Αμήνης θα πρέπει να συντονιστούν στις εσωτερικές πολιτικές με νομοθεσία και να δούμε και ποια είναι τα στρατιωτικά δόγματα και ε, τα σχέδια αντιμετώπισης. Τέλος, να πω δύο λόγια για την προστιθέμενη αξία των ε, κατευθυντηρίων ε, γραμμών. Σέβονται το διεθνές δίκαιο ως έχει και δεν προτείνουν αλλαγές. Ούτε επηρεάζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να περάσουμε σε μια συμπεριφορά που να εξασφαλίζει καλύτερη προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων, ε, ιδιαίτερα ε, στην προστασία τους από τα εμπόλεμα μέρη. Οι κατευθυντήριες γραμμές ε, αφοσιώνονται στο εφικτό. Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και μεγάλα διλήμματα που απαιτούν ρεαλιστικές λύσεις. Υπάρχουν καλές πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούνται στα σχολεία και ε, στα πανεπιστήμια για την προστασία τους. Χρησιμοποιούνται και απευθύνονται σε εμπόλεμες πλευρές. Χρειάζεται τώρα να εφαρμοστούν από ε, ένοπλες ομάδες κρατικές και μη. όλες οι κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να ε, ασχοληθούν με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για να υπάρξει ένας κώδικας ε, για τις ένοπλες φυράξεις. Χαιρόμαστε για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πιο πρόσφατο ψήφισμά σας για τον Νότιο Σουδάν. Ελπίζω να ε, έχουμε την μόνιμη υποστήριξή σας μαζί με τους κρατικούς και μη φορείς, να θαρρύνουμε όλα τα μέλη τα εμπόλεμα να δρουν σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και να τους βοηθήσουμε να το εφαρμόσουν. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η πρόσφατη έγκριση της ε, διακήρυξης για τα ασφαλή σχολεία είναι μια βάση για να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Ήταν μια μεγάλη αφετηρία. Πάνω από 60 κράτη μέλη συμμετείχαν στη διάσκεψη του Όσλο για ασφαλή σχολεία και πάνω από 47 κράτη έχουν τώρα υπογράψει ε, τη διακήρυξη αυτή για τα ασφαλή σχολεία. Ωστόσο, ε, εξακολουθούμε να πιέζουμε όλα τα κράτη να εφαρμόσουν τις ε, κατευθύνες γραμμές και να τα συμπεριλαμβάνουν στα στρατιωτικά τους εγχειρίδια, στις διαταγές, στην εκπαίδευση και στη γενικότερη διάδοση για να ξέρουν σε όλη την ιεραρχία πώς θα χειρίζονται αυτά τα θέματα. Τους επόμενους μήνες η οργάνωσή μας θα βοηθήσει ε, όσο μπορεί για να συμπεριληφθούν αυτές οι ε, κατευθύνες γραμμές στην νομοθεσία, σε εσωτερικές πολιτικές, σε στρατιωτικά δόγματα και σε σχέδια αντιμετώπισης κατεπίγουσων αναγκών. Επίσης, καλούμε την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο μας υποστηρίξει και να συνεχίζει να προωθεί την υλοποίηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. Θέλουμε να καλέσουμε τα κράτη-μέλη που δεν ε, έχουν υπογράψει ακόμα να το πράξουν και να υποστηρίξουν την εφαρμογή τους από τους στρατιωτικούς παντού για να μην γίνουν στρατιωτικές βάσεις τα σχολεία. education in emergency, e Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθηθούν ε, τα σχολεία για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για χώρους μάθησης και όχι για στρατιωτικές βάσεις οι χώρες δωρητές και οι διεθνείς οργανισμοί που δίνουν χρήματα ε, για την ε, παιδεία και για την ασφάλεια θα πρέπει να κάνουν διαβήματα σε χώρες δικαιούχους που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση ή που βγαίνουν από ένα πόλεμο για να εφαρμόσουν αυτόν τον κανόνα για να μην χρησιμοποιούνται στρατιωτικά τα σχολεία. Ε, όλες οι αντάρτικες μη κρατικές ενόπλες ε, ομάδες θα πρέπει να συμπεριλάβουν τις κατευθυντήριες γραμμές ε, στη δράση τους και να καταλάβουν ότι η στρατιωτική χρήση σχολείων και πανεπιστημίων ε, είναι μια κοινή τακτική ε, στον πόλεμο που χρειάζεται μια συντονισμένη απάντηση. Υπάρχουν κανόνες για τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν και κανόνες για τα σχολεία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και χρειάζεται παγκόσμια απόκριση. Όλοι οι μαθητές αξίζουν να είναι σε ασφαλή σχολεία, να φοιτούν ε, και να μπορούν να μαθαίνουν χωρίς φόβο. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν ερώτηση ή να παρέμβουν. Ε, Ευχαριστώ για την παρουσία τους δύο εμπειρογνώμονες και εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντική αυτή η δήλωση για τα ασφαλή σχολεία. Νομίζω ότι η στρατιωτική χρήση των σχολείων είναι κάτι το αρκετά διαδεδομένο, αλλά μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε, πιστεύω. Υπόθηκε και απεδείχθη ότι σε 27 τουλάχιστον χώρες τα σχολεία χρησιμοποιήθηκαν σαν βάσεις, σαν στρατιωτικές μονάδες και από αναγνωρισμένες επίσημες στρατιωτικές ομάδες και από ατάκτους. Είναι μια πρακτική η οποία είναι επικίνδυνη και για τους μαθητές αλλά και για τους διδάσκοντες οι οποίοι θα πρέπει να διακόπτουν λόγω της ανταλλαγής πυρών το σχολείο τους ή και να μην πηγαίνουν διότι θα παραμένουν κλειστά. Εμείς λοιπόν πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε ε, όσο περισσότερες χώρες γίνεται να συνυπογράψουν τις κατευθυντήριες γραμμές. Πρώτον θα πρέπει να ενισχύσουμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση στα πλαίσια των διμερών και πολυμερών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες χρησιμοποιώντας ε, το νέο πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρόλο με τον οποίο οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, μπορέσουν να αναλάβουν δράση στον τομέα αυτό. Επίσης και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι, Νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε το σχολείο σαν κάτι το οποίο διαμορφώνει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. di capire se possiamo impegnare il Parlamento, ma non solo il Parlamento, con una dichiarazione, con una risoluzione, a considerare la scuola come Νομίζω ότι το σχολείο πρέπει να θεωρηθεί σαν ε, κληρονομιά της σύνολης ανθρωπότητας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να θεωρηθεί όπως είπα σαν ανθρώπινη κληρονομιά. Είναι αλήθεια ότι δεν λύνει το πρόβλημα το οποίο έχουμε, αλλά από την άλλη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κυρίως να αναγνωρίζει τη σημασία του δικαίου στην εκπαίδευση και του δικαίου στην παιδική ηλικία. Τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο πάλι στους δύο προσκεκλημένους, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Σράιμπερ που ασχολείται με την προστασία των σχολείων. Ευχαριστώ. Εμείς ε, βλέπουμε πολύ θετικές τις παρουσιάσεις τις οποίες έκαναν οι δύο οργανώσεις. Το ΙΕΣ θεωρεί ότι η προστασία των σχολείων είναι κάτι το κρίσιμο, το βασικό. Εργαζόμεθα με πολλούς τρόπους γύρω από το θέμα αυτό και παρακολουθούμε την ανάπτυξη ε, των κατευθυντηρίων γραμμών της πρότασης για ασφαλή σχολεία ε, το συζητήσαμε και στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Πολλές από τις χώρες μέλη συνυπογράφουν ε, την δήλωση αυτή και τις κατευθυντήριες γραμμές. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση αυτό από κοντά και να καταστήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές ε, δημόσιες ε, και στα πλαίσια της εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των υπαλλήλων που έρχονται αποσπασμένοι από τα κράτη-μέλη. Ζητήσαμε από το Human Rights Watch να παρουσιάσει τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ήταν σημαντική πολύ για μας. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Thank you, uh, thank you, Madam Chair. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Να πω μερικά λόγια μόνο. Το έγγραφο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει οπωσδήποτε περισσότερα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να προσυπογράψουν. Μέχρι τώρα είναι 47, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε η προσπάθεια για να συμβληθούν και άλλες χώρες σε αυτή την κοινή μας προσπάθεια. Έχουμε και μια διαδικασία αναθεώρηση τακτική για να βλέπουμε πώς εφαρμόζονται όλα αυτά και ποιες χώρες εφαρμόζουν τις ε, διακηρύξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές γιατί δεν θέλουμε να μείνει ένα έγγραφο αυτό, θέλουμε να είναι ένα μέσο που να χρησιμοποιείται για πρακτικό τρόπο. Επίσης τονίσατε την σημασία της εκπαίδευσης, παιδείας που είναι βεβαίως και ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και απαραίτητο εργαλείο για την κοινωνική και την ατομική ανάπτυξη. Την περασμένη εβδομάδα στο Όσλο είχαμε μια σύνοδο κορυφή με θέμα την παιδεία για την ανάπτυξη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο και κράτη-μέλη ε, σε πολύ υψηλού επίπεδου εκπροσώπηση και ασχοληθήκαμε με διάφορα ε, θέματα μεταξύ αυτών την εκπαίδευση σε καιρούς και σε περιόδους και χώρες σε ανθρωπιστική κρίση. Το 4% της ε, σύνολης ανθρωπιστικής βοήθειας απευθύνεται στην εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι τα παιδιά ε, περνούν μεγάλο διάστημα σε ε, στρατόπεδα, ε, καταβλισμούς προσφύγων. Δεν είναι για μικρό χρονικό διάστημα εκεί, γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εκπαίδευση από την άφηξή τους και όχι να πούμε καλά βλέπουμε αργότερα τι θα γίνει με το σχολείο. Νομίζω 3% της νορβηγικής ανθρωπιστικής βοήθειας πριν από δύο χρόνια αφιερωνόταν στην παιδεία και αυτό το 3% έχει γίνει σήμερα 8%. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Η κυρία Σάστρε, ευχαριστώ. Το σχόλιο του κυρίου Πανθέρη είναι πάρα πολύ εύστοχο. Για μας το πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που μόλις εγκρίθηκε ένα εξαιρετικό μέσο και εργαλείο θα έλεγα Είναι εξαιρετικό αυτό για να μπορέσουμε να θέσουμε ε, την προοπτική αυτή σε πρακτική εφαρμογή. Περιλαμβάνει κάτι πολύ σημαντικό που είναι η προστασία των παιδιών. Εκεί εστιάζουμε. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα και ο, ο, γνώμονας. Και πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν όλα αυτά. Στα προγράμματα που εμείς εκτελούμε και υλοποιούμε, Πιστεύουμε δεν μπορεί να γίνει σαφής διαχωρισμός, ούτε οφείλει να γίνεται ανάμεσα στα προγράμματα που ε, ε, απευθύνονται στην προστασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση. Το αντίθετο πρέπει να είναι μια συνολική. Όταν μιλούμε για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών χρειάζεται να έχουμε σχολεία και τέτοια κέντρα για να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος προστασίας του παιδιού για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Υπάρχουν και τρόποι ε, να συνδυαστούν τα προγράμματα υγείας και παιδείας και το σχολείο να γίνει ένα ολόκληρο κέντρο, μια κοινότητα, να μην είναι μόνο ε, ε, ένας χώρος εκμάθησης κάποιων και γνώσεων. Είναι μεγάλες οι ανάγκες, το μισό περίπου των αναγκών δεν καλύπτεται παγκοσμίω. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε όραμα δεν είναι μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι προγράμματα προστασίας και βοήθειας στα παιδιά για να μπορούν να εφαρμόζονται και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με την πρόταση που κάνετε. Τα σχολεία να κηρυχθούν σε παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας. Όλα τα σχολεία. Αυτό είναι θέμα των κυβερνήσεων. Εμείς αυτό που θέλουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης όλων των παιδιών είναι μια ευκαιρία για να έχουν μια καλύτερη ζωή και στο παρόν και στο μέλλον. Να βελτιώνουν τη ζωή τους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία στην οποία είναι μέλη. Έχω κι εγώ ένα σχόλιο. Προηγουμένως το συζήτησα με τον Υπουργό και είναι αυτό που έχει να κάνει με την ανυπαρξία σχολείων. Δηλαδή το σχολείο, ε, μιλάμε για το σχολείο ως ένα ασφαλή ε, τόπο, ένα ασφαλές καταφύγιο. Αλλά στα στρατόπεδα, καταβλισμούς προσφύγων, πολλές φορές δεν υπάρχει καθόλου σχολείο. Και περνάνε ολόκληρες γενιές εκεί παιδιών τη ζωή τους. Αυτό πώς θα το λύσουμε, πώς θα εντάξουμε τα ασφαλή σχολεία ε, σε τόπους που πολλές φορές δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν χώροι ε, με μια στοιχειώδη ηρεμία για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν κάτι για τη ζωή τους. Θα μπορούσαμε κάπως να το αναφέρουμε στη συζήτηση και αυτό το θέμα. Τι να κάνουμε για να μπορέσουν τα κορίτσια και τα γόρια να έχουν ασφαλή τόπους να μαθαίνουν και πέρα από το καθεστώς του πρόσφυγα να μορφώνονται και να μην διαιωνίζεται αυτό το καθεστώς. Yo Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ε, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. Αν υλοποιήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε για αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που μεγαλώνουν ε, εκτοπισμένα σε καταβλισμούς προσφύγων, σε κέντρα μακριά από τα σπίτια τους και επιπλέον υπάρχουν παιδιά που ζουν σε κοινότητες, σε, σε χώρες υποδοχής που δεν είναι καν καταγεγραμμένα και δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Ή όταν πηγαίνουν υφίστανται τεράστιες πιέσεις. Ας πούμε τη, σύγκρουση, τη σύραξη στην Συρία υφίστανται τεράστιες πιέσεις και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το κάθε παιδί. και τα παιδιά της χώρας υποδοχής και τα παιδιά πρόσφυγες. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι πολλά παιδιά σήμερα δεν ε, μένουν λίγο διάστημα σε προσφυγικούς καταφλισμούς αλλά όλοι τους στην παιδική ηλικία. 37 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία λόγω των σειράξεων ενώ 59 εκατομμύρια συνολικά στον κόσμο δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Αν δεν ασχοληθούμε με το θέμα της παιδείας σε σειράξεις και υπάρχει κίνδυνο σε πολλά μέρη του κόσμου να χαθεί μια γενιά και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας και για το έργο σας γενικότερα. Θα σας ε, συνοδεύουμε, θα σας πλαισιώνουμε με διάφορους τρόπους. Ε, θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Το πρώτο που σκεφτήκαμε είναι να κάνουμε ερώτηση στο Συμβούλιο για το πώς ενέχονται τα κράτη-μέλη που ακόμα δεν έχουν προσυπογράψει σε αυτή την προσπάθεια τις κατευθυντές γραμμές τους ερχόμενους μήνες. Δηλαδή από τη δική μας Επιτροπή θα δώσουμε συνέχεια και θα παρακολουθούμε την εργασία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθατε. vamos a Το επόμενο θέμα είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη. Υπήρξε ένα ψήφισμα την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρώτα θα είχαμε συζητήσει το θέμα για την κατάσταση στην Καμπότζη και θέλω να υπογραμμίσω εδώ την παρουσία του Γκαέλ Ντουσελ και του Δόκτωρα Κέκ. Θα μας μιλήσει για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη και έχει το λόγο πρώτη η κυρία Κέκ. Νομίζω ότι είναι το μικρό σας όνομα. Vous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 γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιόν σας σήμερα. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για το ψήφισμα που δεχτήκατε για τη σοβαρή απειλή που αντιπροσωπεύει στην ελευθερία ε, έκφρασης η κατάσταση στην Καμπότζη. Οι ανησυχίε σας είναι δικαιολογημένες στο μέλλον. Το νομοσχέδιο για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα αποτελεί επιτρέψει, θα απαγορεύει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να κάνουν δηλώσεις για την Καμπότζη. Και ψηφίστηκε χωρίς την αντιπολίτευση, τη απουσία της αντιπολίτευσης. Ο λόγος είναι απλός. Τα κριτήρια για την εγγραφή στα μητρώα των οργανώσεων κρίνονται από την εθνική ασφάλεια. Παραδόσεις, η δημόσια τάξη και η πολιτική ουδετερότητα ανοίγουν το δρόμο για οποιαδήποτε αυθαίρετη απόφαση απαγόρευσης οργανώσεων. Είναι λοιπόν απαραίτητο να θυμηθούμε ότι η κοινωνία των πολιτών δεν είναι εχθρός της κυβέρνησης ή του καμποτζιανού λαού αλλά ουσιώδης εταίρος στον διάλογο μεταξύ του εκτελεστικού και της κοινωνίας και θα έπρεπε να είναι επίσης ουσιώδης εταίρος για οποιαδήποτε κοινωνική και οικονομική αναπτυξιακή πολιτική. Γι' αυτόν τον λόγο η δραστική μείωση της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης έκφρασης θα ήταν πολύ αρνητική πολιτική κίνηση. Εκτός αυτού, λόγω του υπάρχοντος συντάγματος του αστικού κώδικα και του ποινικού κώδικα, η Λάγκο δεν είναι μόνο άχρηστη κατά αυτού, αλλά και μη συνταγματική. Παραβιάζει τα, τις συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Σύνταγμα, καθώς και την, συμφωνία, Συμφωνία των Παρισίων που υπέγραψαν τα τέσσερα καμποτζιανά κόμματα τον Οκτώβριο του 1991 με 18 χώρες και με μάρτυρα τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ε. Τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα που εγκρίθηκε και από την Καμπότζη το 1992 και το Σύνταγμα της Καμπότζης του 1993 που δηλώνει ότι το Βασίλειο σέβεται όλες τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων άρθρο 31, 41 και 42 του Το λάγκο είναι άχρηστο εφόσον ο ποινικό κώδικας, ο αστικός κώδικας, η, τα νομοσχέδια κατά της τρομοκρατίας και της διαφθοράς όλα ισχύουν και αρκούν για να εφαρμοστούν οι κανόνες που αφορούν τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλες οργανώσεις. Είναι αρνητικό διότι θα αποτρέψει κάθε θετική εισφορά από την κοινωνία των πολιτών για την πιο αρμονική και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Εδώ παραδείγματα του αρνητικού του χαρακτήρα. Πρώτον, το Λάγκο επιβάλλει υποχρεωτική εγγραφή για όλες τις τοπικές και διεθνείς οργανώσεις και μη κυβερνητικές διάφτες. Βέβαια η λέξη που χρησιμοποιείται association μπορεί να αφορά οποιονδήποτε μέχρι και τεράστιες διεθνείς οργανώσεις. Το, το Υπουργείο Εσωτερικών, ΙΠΕΣ, έχει απόλυτη δικαιοδοσία για να εγκρίνει ή να απορρίψει την εγγραφή. Και άρα θα γίνεται με πολιτικά κριτήρια η εγγραφή μπορεί να τύχει άρνησης με, για λόγους που λένε ότι μπορεί η οργάνωση αυτή να εμπαρεμποδίσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δημόσια τάξη ή να βλάψει την εθνική ασφάλεια και, λοιπά, και τις παραδόσεις της καμποζιανής κοινωνίας. Το Λάγκο απαγορεύει οποιαδήποτε δραστηριότητα των μη εγγεγραμμένων οργανώσεων με πρόστιμο πάνω από 10 εκατομμύρια ριάλ ή 1220 με 2.440 αμερικανικά δολάρια ή μπορεί και να διωχθεί ποινικά. Τέταρτον, δεν υπάρχει πρόσβαση σε κανένα νομοθετικό μέσο. Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής. Πέμπτον, αφού δραφούν όλες οι διεθνείς και τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν την υποχρέωση να διατηρούν πολιτική ουδετερότητα όπως λένε. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τη ρήτρα αυτή για να διαγράψει οποιαδήποτε οργάνωση που ασκεί κριτική. Έκτον, η νέα μορφή δεν επιτρέπει θεωρητικά την επανεγγραφή μιας οργάνωσης αφού έχει διαγραφεί. Αυτό είναι καινούριο. Έβδομον, το Λάγκο χορηγεί τη δικαιοδοσία στην κυβέρνηση να σταματάει να κόβει τις σχέσεις με διεθνείς οργανώσεις και να διώκει, να διώχνει από τη χώρα εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων. Τέλος, υπάρχουν αυστηρές διατάξεις που δίνουν το δικαίωμα στην κυβέρνηση να ελέγχει τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση των κοιόμικρων καθώς και να επιβάλλει αλλαγή της ηγεσία τους. Συμπέρασμα σήμερα η Καμπότζη έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Σχεδόν 25 χρόνια μετά τη Συμφωνία των Παρισίων που αποτελούσε το τέλος 11 χρόνων βιετναμέζικης κατοχής και πάνω από 20 χρόνια εμφυλίου με τρομερές τραγωδίες που κατέστρεψαν στους ανθρώπινους πόρους στην Καμπότζη καθώς και την τεχνογνωσία υπάρχουν ακόμη. Τα πολιτικά κόμματα διαπράττουν, ε, εφαρμόζουν έναν ήθη διαλόγου αλλά απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε αυτό οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Ενώ οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα του διαλόγου και να βελτιώσουν την πολιτική αρμονία του Βασιλείου. Στον, στον 21ο αιώνα όπου είναι πια αδύνατο να διοικηθεί μια χώρα χωρίς τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών η καταστροφή της δυνατότητας θετικής κριτικής, επικοδομητικής κριτικής είναι η παναχώρηση και στρώνει το δρόμο για νέες εντάσεις με τους αγρότες, τους εργάτες, τους δημοσίους υπαλλήλους, την νεολαία, τους κοινοτικούς ηγέτες, ακόμη και τους βουτιστές μοναχούς. Και επίσης δημιουργεί καχυποψία και ρίχνει μια σκιά στην αληθινή πρόθεση της ηγεσία της Καμπότζης. Αφού η κοινωνία των πολιτών και η κυβέρνηση και οι δύο στοχεύουν στο ίδιο πράγμα, αρμονική ανάπτυξη θα έπρεπε να συνεργάζονται και να μην θεωρούν ο ένας εχθρό τον άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντιουσεπίλκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Για 10 λεπτά. Η FDR συμμερίζεται τις απόψεις που εξέφρασε η προλαλή Τα θέματα τα οποία τίθενται με το νέο νόμο ο οποίος έγινε δεκτός, το δικαίωμα του συνέρχεστε και ο νόμος για τα μήκυο, θέτει ένα πρόβλημα το οποίο έχει καταγγελθεί ομόφωνα από το σύνολο των διεθνών ΜΚΟ και των τοπικών Καμποτζιανών ΜΚΟ, όπως επίσης και των εμπειρογνωμόνων. Euh, euh, Νομίζω ότι αυτή η νέα νομοθεσία είναι αντίθετη με το σύνολο των διεθνών επιπέδων και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα που έχει επικυρώσει και η ίδια η Καμπότζη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε και αυτή εδώ και πολύ καιρό ασχολείται με τα θέματα αυτά ήδη από το 2008. Παρενέβη λοιπόν και στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ομιμοποίηση του ρόλου των ΜΚΙΟ στις διάφορες χώρες. Ανταποκρίνεται στο σύνολο των κατευθυντηρίων γραμμών και στην παρουσία της νομοθεσίας γύρω από τα θέματα αυτά στη διεθνή σκηνή. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τους κινδύνους που δημιουργεί για το μέλλον ο νόμος αυτός και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος αυτός θα φέρει περισσότερα εμπόδια στο σύνολο των θεμάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Καμπότζη. Το θέμα των παράνομων κρατήσεων, το θέμα της διαφοράς, το θέμα της σωστής διακυβέρνησης, της ανεξαρτησίας ε, της δικαστικής εξουσίας, όλα αυτά ε, όπως και οι κατασχέσεις γεών, ο νέος νόμος για τους συλλόγους, ενώσεις και οργανώσεις δημιουργούνται προβλήματα στην καθημερινή μάχη η οποία έχει οξυνθεί λόγω των κατασχέσεων γεών και των πιέσεων και της κατασχολής εις βάρος των πρασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν υπάρξει επίσης και πάρα πολλές ενέργειες εις βάρος ε, της άλλης ένωσης, της ΑΝΤΟΚ που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα πλαίσια πάντα διαδικασιών κατασχέσεως γεών. η ΑΝΤΟΚ και η δική μας οργάνωση ελέγχονται σε επίπεδο δικαστικό και διοικητικό διότι έχουν πιέσει τη δικαστική εξουσία και δήθεν έχουν κατασυκοφαντήσει επειδή καταδίκασαν τη σύλληψη και καταδίκη δύο χωρικών στα πλαίσια μιας διαφοράς για την κατάσχεση γεών. Όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πράγματι να συνεχίσει ε, την πορεία και την πολιτική της απέναντι στην Καμπότζη, πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά όλα αυτά τα προβλήματα και να συνεχίσει να πιέζει, να συνεχίσει να ανακοινεί τα διάφορα προβλήματα και να πολλαπλασιάζει τα μέσα παρέμβασης. Για το θέμα της κατάσχεσης γεών, για αναγκαστικής απαλωτρίωσης, το θέμα αυτό δεν έχει επιληθεί ακόμα. Η Αλικαντό έδωσε τεκμήρια σύμφωνα με τα οποία υπήρξαν άλλα 108 προβλήματα ε, που έφυξαν χιλιάδες οικογένειες. Στα πλαίσια της δικής μας οργάνωσης εμείς έχουμε ασχοληθεί με δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις στον τομέα της παραγωγής σαχαροκαλάμου και στον τομέα παραγωγής καουτσούκ. Τα δύο θέματα αυτά δεν έχουν επιληθεί ακόμα Έχουμε αποστείλει πρόσφατα μια ανοιχτή επιστολή, ε, ίσως και να την έχετε διαβάσει. Λοιπόν τώρα συστάσεις για τη συνέχεια. Εμείς θέλουμε στο μέλλον να κρατήσουμε ανοιχτό το θέμα της Καμπότζης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. να λάβουμε υπόψη μας τις επόμενες σημαντικές ημερομηνίε τον μήνα Σεπτέμβριο στα Ηνωμένα Έθνη, Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ζητάμε να υπάρξει μια σκληρή γλώσσα για τις παραβιάσεις στον τομέα της ελευθερίας έκφρασης κτλ. και για τα θέματα των απαλωτριώσεων. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια ανανέωση και της εντολής του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση καλύτερα. Τώρα, μια δεύτερη χρονική προθεσμία σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι το λεγόμενο shrinking space. Αυτό αφορά την επικράτηση χρηστών πρακτικών και εδώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια συνάντηση τον μήνα Δεκέμβριο και θα οργανωθεί από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και θα έχει σαν στόχο τη διασύνδεση ανάμεσα στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το λεγόμενο shrinking space, τον συρρυκνούμενο χώρο ή το συρρυκνούμενο διάστημα. Μια καλύτερη μορφή συντονισμού της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και του Κοινοβουλίου θα αποδείξει ακριβώς τις χρηστές πρακτικές, τις αποτυχίες και τις δυσκολίες τις οποίες είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και τέλος, και τελειώνω, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί θέτοντας ε, ε, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για δύο βασικά θέματα, το γιατί σε ανώτερο επίπεδο δεν ακούγονται δημόσια θέσεις ε, γύρω από το νόμο αυτό και δεύτερον για τον τρόπο με τον οποίο στο μέλλον θα τηρήσουμε μια διαφορετική στάση στα θέματα της ανάπτυξης απέναντι σε τέτοιες χώρες, ενισχύοντας τους τοπικούς πληθυσμούς που είναι πιο ευάλωτοι και στον τομέα των διαφορών ε, επί των γεών και βοηθώντας την κοινωνία των πολιτών για την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, στην Καμπότζη και μετά θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, έτσι, ε, με πιάσετε λίγο εξαπίνης, δεν ήξερα ότι θα μου δίνατε το λόγο. θα ήθελα να συμπληρώσω σύντομα μερικά πράγματα στις δύο παρεμβάσεις. Σε ό,τι αφορά για τον νόμο για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα σωματεία, ομολογώ ότι προσωπικά έχω κάπως απογοητευτεί από το γεγονός ότι τόσο γρήγορα εγκρίθηκε αυτός ο νόμος. Εργαστήκαμε πάρα πολύ από αυτού εδώ και πάρα πολλά χρόνια όπως υπόθηκε και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες ήμασταν σε πάρα πολύ στενή επαφή με τους εταίρους μας και με την κυβέρνηση και θα επιθυμούσαμε να είχαν ε, επεξεργαστεί περισσότερο μαζί μας κάποια στοιχεία για να ε, μην ε, περνούσε τόσο βιαστικά όπως είπε η Δόκτωρ Κέκ. Τώρα όλα είναι ζήτημα ερμηνείας αυτού του νόμου και πώς θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση. Ένα σημαντικό για μένα ζήτημα θα ήθελα να αναφέρω και θα πρέπει κάπου να αναφέρεται. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που τώρα είναι ε, εγγεγραμμένες στην Καμπότζη, διεθνείς ή εθνικές, ε, παραμένουν καταχωρισμένες. Δεν χρειάζεται νέο μητρό. Βεβαίως μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να ε, διαγραφούν με το νέο νόμο, αλλά δεν χρειάζεται ε, από την αρχή εγγραφή η νέα καταχώρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει διαβήματα με τα κράτη-μέλη επιτόπου, με τις αντιπροσωπείς και τις πρεσβείες για να ελέγχουμε προσεκτικά και να παρακολουθούμε οποιαδήποτε καταχρηστική θα έλεγα ερμηνεία του νόμου. Ε, επίσης, σε ό,τι αφορά τα θέματα της χρήσης γης, ε, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και την αντιπροσωπεία στο, στην Καμπότζη είναι προτεραιότητα. Ίσως υπαριθμόν ένα θα έλεγα στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη χώρα αυτή. Σε τρία επίπεδα είναι η δράση μας και η παρέμβασή μας. Πιο διαρθρωμένη, δηλαδή έχουμε πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση και τους αναπτυξιακούς εταίρους για τα θέματα αυτά των γεών και αναφέρει τακτικά η κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται και πώς εφαρμόζουν μια οδηγία που εγκρίνανε τον Μάιο του 2012 για τη βελτίωση της ε, κατάστασης ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας γεών και ε, τις ε, περίφημες παραχωρήσεις οικονομικές των γεών ε, που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση. Τις τρεις τελευταίες χρονιές είχαμε ένα διάλογο για αυτά τα θέματα, για την αναθεώρηση των παραχωρήσεων, για τη χορήγηση τίτλων ιδιοκτησίας. Κάποιες συμβάσεις διακόψαν, σταμάτησαν, συνεχίστηκαν και θα υπάρξει μια διανομή ε, με κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, αναφερθήκατε ιδιαίτερα για γεγές ε, όπου καλλιεργείται ζάχαρο Έχω ασχοληθεί και με έχει απασχολήσει πάρα πολύ όσο και ανησυχήσει αυτό το θέμα ε, κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Καμπότζη. Υπήρξαν πρόοδοι, ακόμα και αν δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Δημιουργήθηκε μια διυπουργική ε, ομάδα εργασίας η οποία θα επιφορτιστεί με το έργο να δει έναν τρόπο να αντισταθμιστούν, να αποζημιωθούν οι οικογένειες και οι κοινότητες που έχουν ε, πληγεί από αυτές τις απολυτριώσεις για την καλλιέργεια ζαχαροκαλάμου. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση για να αρχίσει ένας λογιστικός έλεγχος των ε, διεκδικήσεων που προβάλλουν οικειό, κοινότητες τοπικές και οικογένειες. Και ένα τελευταίο θέμα, τρίτο, στο Ευρωπαϊκό Μέσο για την Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μία από τις προτεραιότητες που ήταν και παραμένει βασική στη βοήθειά μας, είναι βεβαίως οτιδήποτε έχει να κάνει ε, με τις διενέξεις και τις διαφορές για θέματα γεών. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα Θέλω να πω στους παρόντες βουλευτές ότι στην Καμπότζη μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους μας εταίρους, τα κράτη-μέλη δηλαδή, και την Ελβετία επίσης, έχουμε αναπτύξει μια κοινή στρατηγική αναπτυξιακή συνεργασίας με την Καμπότζη. Με κεντρική ιδέα ακριβώς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση, και θεωρούμε ότι θα είναι ενδιαφέρον και σημαντικό εργαλείο για τον πολιτικό διάλογο που θα έχουμε την Καμπότζη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Ροτμπίλερ. Λοχ Μπίλερ. Όχι, Ροτ The... Ευχαριστώ και για τις συστάσεις που κάνατε και για την περιγραφή της κατάστασης. Έχω όμως ορισμένες απορίες για να το δω. Λοιπόν, τόσο από το Λάγκο που πέρασε χθες. Ανακοινώνονται και μελλοντικά νομοσχέδια για τα συνδικάτα και για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Μου φαίνεται απριόριο ότι αυτά τα δύο νομοσχέδια βασικά θα υπονομεύσουν και αυτά δημοκρατικά κριτήρια και πρότυπα. Πώς το βλέπετε αυτό και μπορεί να υπάρξει χειροτέρευση των δημοκρατικών δομών στην Καμπότζη και όπως είπατε δόκτωρα που, είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς πόσο ενεργή κοινωνία των πολιτών υπάρχει στην Καμπότζη. Είπατε και εσείς ότι ο στόχος πρέπει να είναι η κυβέρνηση να συμβαδίζει με τις, να δέχεται και τις επικρίσεις και τις συστάσεις της κοινωνίας των πολιτών για να αναπτυχθεί περισσότερο η κοινωνία. Είναι λοιπόν λυπηρό ότι με όλα, όλες τις παρεμβάσεις ε, που γίνονται από την Ένωση μερικές χώρες μέλη και το κοινοβούλιο μας τις περισσότερες φορές δεν έχουν ακουστεί αυτά τα μηνύματα που είναι επικίνδυνα για τον περιορισμό της λειτουργίας των μήκη όμικρον. Τώρα η κυρία Ντουσεπούλκρ μας είπατε και για το άλλο νομοσχέδιο που θα δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς για το νομοσχέδιο δηλαδή για την ένομη τάξη. Ήδη διαβάζω ότι η Διεθνής Οργάνωση για την Ένωμη έχει χειροτερεύσει το καθεστώς της Καμπότζης γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει λογοδοσία για θανάσιμους πυροβολισμούς κατά εργαζομένων στην υφαντουργία και δεν έγινε και καμία έρευνα για τη δολοφονία ανθρώπων που ασχολούνταν με την προστασία του περιβάλλοντος. Ούτε καμία δίκη. Ήδη λοιπόν υπάρχουν θέματα εδώ για την ερμηνεία της έννοιας της ένομης τάξιος. Και πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό όταν μιλάμε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη. Τώρα, μια και είναι εδώ ο πρεσβευτής Κότα, έμαθα από εσά ότι και στην Πνόμ Πεν χορηγούνται γέες για φυτίες ζαχαροκάλαμου που ανήκουν σε μια ενωσιακή εταιρεία και λειτουργούν με συνθήκες δουλοκτησίας. Ίσως το κοινοβούλιο μας θα έπρεπε να σκεφτεί μήπως θα έπρεπε να ενδυναμώσει τις σχέσεις του με το Καμποτζιανό Κοινοβούλιο στο μέλλον, στο μέλλον όχι αμέσως να έχουμε πιο στεναρές σχέσεις Μάλιστα ε, Θέλετε να απαντήσετε πρώτα κύριε Πρέσβη και μετά θα δώσω το λόγο στις κυρίες σας Ευχαριστώ. Στα αγγλικά. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση σας για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία που ενέχεται στην ε, παραχώρηση για το ζαχαροκάλαμο. Δεν είναι ευρωπαϊκή, αμερικανική είναι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, εκκρεμεί στη δικαιοσύνη μια υπόθεση σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, σε ένα, ενός κράτους μέλους. Υπάρχει και εξωδικαστική επίλυση. Προσπαθούν να βρουν ένα συμβασμό ε, εκτός δικαστηρίου και χρειάζεται μια εξωτερική ε, λογιστική παρακολούθηση με τον λογιστικό έλεγχο που αρχίζει όπως είπαμε τώρα και αφορά και τη συγκεκριμένη παραχώρηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαλαμπρού. Ε, thank you, Σας ευχαριστώ κυρία μου που με ρωτήσατε για τον νόμο μετά το Λάγκο, δηλαδή τι μέλη γενέστε. Χθε η κυβέρνηση ενέκρινε στην Εθνοσυνέλευση το νόμο αυτό, απουσία της αντιπολίτευσης. Στην Εθνοσυνέλευση μας είναι δύο τα βασικά κόμματα, η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Αυτά. Το ΣΕΝΑΠΗ που λέγεται το κόμμα της αντιπολίτευσης ε, ε, μποϊκοτάρει το κοινοβούλιο και δεν μετέχει. Οπότε ένα κόμμα ενέκρινε αυτό το νόμο. Είναι γεγονός αυτό που είπατε. Ε, έχουν τρία νομοσχέδια, τώρα ένα για τα συνδικάτα, για το συνεταιρίζεστε που είναι πάρα πολύ περιοριστικός ο νόμος για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί, να συσταθεί ένα συνδικάτο. Μέχρι σήμερα δεν χρειάζεται άδεια του Υπουργείου Εργασίας. το εξή όμως, εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο και γίνει νόμος, για να λειτουργήσει μια συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει να ζητήσει την άδεια του Υπουργού Εργασίας. Και 20% των ε, εργαζομένων πρέπει να είναι μέλη για να δημιουργηθεί ένα συνδικάτο. Και αν θέλουν να κάνουν μια ομοσπονδία συνδικάτων, πρέπει να συγκεντρώνουν 15 συνδικαλιστικές οργανώσεις για να συνασπιστούν και να γίνει ομοσπονδία. Ενώ για την συνομοσπονδία χρειάζονται 10 ομοσπονδίες. Οπότε είναι υπερβολική η περιορισμοί για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Και επίσης, μπορεί η κυβέρνηση να τους αναγκάσουν να πληρώσουν πολύ υψηλά τέλη τώρα η εισφορά των μελών ε, είναι κάτι στο οποίο εναπόκειται στο συνδικάτο να το ορίσει, ανάλογα με τους χαμηλούς μισθούς των εργαζομένων. Ε, τώρα, αν έρθει το κράτος να θεσπίσει υποχρεωτική εισφορά ενό ύψους, θα είναι πολύ κακό. Ε, μιλήσατε για μια δολοφονία, ε, ότι δεν ακολούθησαν έρευνες. Από το 1994 ήταν πολύ, όχι μόνο ο κύριος ο συγκεκριμένος. Από το 1994 μέχρι το 2012 δολοφονήθηκαν 12 δημοσιογράφοι μέρα μεσημέρι ε, με μαφιόζικο τρόπο και ο δράστης προσήχθη στη δικαιοσύνη. και τρεις συνδικαλιστές όπως ο κύριος ε, που αναφέρατε δολοφονήθηκαν πάρα πολύ γνωστοί χωρίς έρευνα, περαιτέρω και δίωξη. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επανέρχομαι στους νόμους για τις τηλεπικοινωνίες, για το έγκλημα στο κυβερνοφόρο, ε, χώρο, συγγνώμη. Και για τη Γεωργία, αν περάσουν αυτοί οι τρεις νόμοι, τότε θα νομιμοποιηθούν όλες οι παραχωρήσεις γεών. Έχουμε τέτοια προβλήματα στην Καβότζη και επίσης μιλήσατε και για πυροβολισμούς, ε, για την καταστολή ε, των εργαζομένων στις αρχές του Ιανουαρίου του 2014. Ναι, όντως. Διαδήλωναν μπροστά στο εργοστάσιο οι εργάτες και ζητούσαν αύξηση του μισθού τους. 177 δολάρια παίρνουν που είναι ο ελάχιστος μισθός. Ο κατώτατο. Ε, δεν ζει κανεί. έστω και ε, ένα άτομο είναι στην Πνομπέχ. Λόγω του πληθωρισμού. Ζητούν λοιπόν αύξηση του κατώτατου μισθού και επίσης πιο αξιοπρέπει συνθήκες εργασίας. Και κατέβηκε η στρατιωτική αστυνομία και τους πυροβόλησε με πέντε νεκρούς, έναν αγνοούμενο και 40 τραυματίες. Ορισμένοι ήταν πάρα πολύ σοβαρά τραυματίες. Το γνωρίζουμε γιατί εμείς τους περιθάλψαμε αυτούς τους 40. Και επίσης ε, συνέλαβαν 23 χωρίς ένταλμα σύλληψεως. Τους ε, κράτησαν σε ένα ε, μέρος που είναι πάρα πολύ μακριά για τις οικογένειές τους, στα σύνορα με το Βιετνάμ, που έχουμε μια φυλακή που ονομάζεται CC3, εκεί ε, ε, κρατήθηκαν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους επισκεφθούν οι οικογένειές τους. Αυτά. Έτσι έχει η κατάσταση λοιπόν στην Καμπότζη. Η ατιμορρησία οργιάζει και το κράτος δικαίου επίσης. Ε, είναι προβληματικό, είναι κάτι που μας απασχολεί. Πριν δώσω το λόγο τώρα στην κυρία του Σερπίλκ, ζήτησε ο κύριος Παντζέρη το λόγο. Ένα μικρό σχόλιο. Ήδη το να λέει κανείς ότι δεν έχει νόημα το να έρθει εδώ κάποιος να κάνει δηλώσεις αυτό δηλεί μια μη δημοκρατική χώρα. Ο Πρωθυπουργό Σεν συμπληρώνει παρουσία 30 ετών περίπου στην εξουσία. Πέρα από αυτό, το οποίο εμένα μου δημιουργεί μια κάποια αλλεργία βέβαια, αλλά πες ότι αυτό είναι προσωπική μου αντίληψη. Πρέπει να πω ότι από ό,τι άκουσα και από ό,τι γνωρίζω έχουμε να κάνουμε στην Καμπότζη με, μια, με ένα πολιτισμό βίας και ατιμορρησίας. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα της Καμπότζης. Έχουμε περάσει ένα ψήφισμα εμείς, αλλά υπάρχει η άποψη βέβαια στην κοινή γνώμη την ευρωπαϊκή ότι υπήρχε η τραγωδία των Ερυθρών Χμέρ αλλά ό,τι ακολούθησε μετά είναι αναγκαστικά και υποχρεωτικά καλύτερο. Λοιπόν, πρώτον παρατήρηση ακολουθείται από μια ερώτηση. Καταρχάς, θα πρέπει να περιμένουμε την ερμηνεία για το νόμο αυτό, για τις διάφορες οργανώσεις. Γιατί όπως είπα, είμαστε την παρουσία μιας κουλτούρας βίας και ατιμορρησίας. Οπότε ο νόμος αυτός δυστυχώς θα περιορίζει τις δυνατότητες των μικιών και τις δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών να εκφραστεί ελεύθερα. Πολύ σωστά λοιπόν, όπως υπόθηκε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία στήριξης αυτών που αμφισβητούν τον νόμο. Δεύτερη παρατήρηση ερώτηση. Υπάρχει αντιπολίτευση στην Καμπότζη. Αυτά τα οποία βλέπω όμως είναι ότι στην ουσία δημιουργείται ένα μοναδικό κόμμα την Καμπότζη εξουσίας και αυτό είναι περιοριστικό, περιοριστικό συγγνώμη, για τη δημοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντουισεπίλκρ θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Η ε, ερώτηση την ξέχασα. Μου διέφυγε. Του κυρίου Παντζέρη για το ενιαίο κόμμα, για το μοναδικό κόμμα. Ε, ναι, Για την αναγκαιότητα να μην περιμένουμε την ερμηνεία του κράτους. Πράγματι, όπως σας είπα, η νομοθεσία αντιβαίνει με τα διεθνή πρότυπα γιατί είναι πολύ ασαφής και η ασάφεια αυτή έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για αυθαίρετες κρατήσεις. Ασαφής εννοώ ότι δεν συμφωνεί με κανένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο για να ξέρει κανείς τι να αναμένει. Διότι η νομοθεσία δεν εφαρμόζει τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας για να ανταποκριθούμε στο αδίκημα που προσάπτουν ούτε προβλέπονται σαφώς οι κυρώσεις. Νομίζω ότι απαντήσαμε πλήρως στο θέμα του κράτους δικαίου ήδη. Για μας είναι ουσιώδες θέμα η δυνατότητα να συνδεθεί η ελευθερωτική ελεύθερη έκφραση με το κράτος δικαίου είναι κάτι που το στηρίζει η Ένωση γιατί όμως στηρίζει και την Καμπότζη γιατί έχει πολλά προγράμματα αναπτυξιακά. Όσο για αυτά που είπε ο κύριος Κοτάν θα ήθελα να πω ότι για τη διαδικασία που εφαρμόστηκε και το μορατόριο του 12 το θέμα της διαφάνειας των διομολογήσεων ε, δεν έχει ακόμα λυθεί. Μπορούν και τώρα να δοθούν διομολογήσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσει να ενδιαφέρεται γι' αυτό η Ένωση έπειτα. Ε, ε, για τη ζάχαρη εδώ παραμένουν ακόμη πολλά ανοιχτά θέματα γιατί όπως είπατε θα εξεταστούν τώρα τα φυτά αλλά τα ζαχαροκάλαμα δηλαδή αλλά δεν είναι γνωστό πώς θα υπολογιστούν οι αποζημιώσεις και οι καθαρά παράνομες εκχωρήσεις ή διομολογήσεις που δόθηκαν τι θα γίνουν θα επιστροφεί η γη στα άτομα από τα οποία την πήραν. Και τελικά η νέα νομοθεσία τελικά τα θέτει όλα αυτά εν κίνδυνα. Εσείς με το μαλλί. Ε, ρωτήσατε αν η Καμπότζη έχει μονοκομματικό σύστημα. Υπάρχουν δύο κόμματα, υπάρχει αντιπολίτευση στη Βουλή. Παρόλα αυτά, όλα τα νομοσχέδια που έχουν περάσει απαιτούν απλώς 50 συν 1 πλειοψηφία. Άρα δεν μετράει η άποψη της πλειοψηφίας les 55 membres de l'opposition ne se sont pas Και μερικέ φορέ η αντιπολίτευση μποϊκοτάρισε την ψηφοφορία, αλλά παρόλα αυτά πέρασαν οι νόμοι. Πέρασαν επίση τρία νομοσχέδια για τον έλεγχο του δικαστικού χωρί παρουσία της αντιπολίτευση και τα τρία αυτά νομοσχέδια έλεγαν ότι το εκτελεστικό, η κυβέρνηση ελέγχει το δικαστικό τομέα. Δεν υπάρχει λοιπόν διαχωρισμός των εξουσιών στην Καμπότζη, όπως αντίθετα το προβλέπει το Σύνταγμα. Η νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία ελέγχονται όλα από το κυβερνών κόμμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως η τηλεόραση. Σχεδόν όλα τα κανάλια ελέγχονται από το κυβερνών κόμμα. και αν πρόκειται να δοθεί άδεια σε μια ιδιωτική εταιρεία για να μπορούν να εκφραστούν εκεί η αντιπολίτευση και η μήκη ο μικρόν μια ανεξάρτητη τηλεόραση δηλαδή αυτό είναι πολύ δύσκολο δυσκολεύεται η αντιπολίτευση να βρει τα τρία εκατομμύρια που απαιτούνται γι' αυτό δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα είναι λοιπόν πολύ δύσκολο στην Καμπότζη να μιλήσει κανείς για πολυκομματισμό όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Υπάρχουν δύο κόμματα ε, seulement d'un parti politique. αλλά μόνο το ένα άδρα. Και μια τροποποίηση του Συντάγματος θα απαιτούσε πλειοψηφία δύο τρίτων. Η δε ψήφος εμπιστοσύνης απαιτεί απλώς 51%. Το ΠΠΣ λοιπόν θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει και γι' αυτό φοβόμαστε. Νομίζουμε ότι ο κίνδυνος να ψηφιστεί ο νόμος για τα συνδικάτα, για το κυβερνοέγκλημα, για τη γεωργία, όλα αυτά μπορεί να ψηφιστούν μόνο από το κυβερνών κόμμα. Pour les foncières, je suis d'accord avec αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα τελικά γιατί μπορεί κανείς να πει ότι 63% του καλλιεργήσιμων γεών έχουν δοθεί χαριστικά σχεδόν στις ιδιωτικές εταιρείε και πάνω από 700.000 Καμποτζιανών έχασαν τη γη τους, εκδιώχτηκαν από τη γη τους. Λέγεται relocation site εκεί που τους πάνε αλλά πρέπει να δείτε πώς είναι χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς σχολείο εκεί κοντά για τα παιδιά, χωρίς σέλτερ, τίποτα. Ούτε job. Είναι κάτι αλάνες που δίνουν στον κόσμο που ζουν πια σαν πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Και γι' αυτό πολλοί από αυτούς φεύγουν για να ψάξουν δουλειά εκτός της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδων πηγαίνουν στην Ταϊλάνδη, στη Μαλαισία και στην Νότια Κορέα. Πολλοί Καμποτζιανοί. Μερικά, σε μερικά χωριά βρίσκει κανείς μόνο πολύ νέους ή πολύ ηλικιωμένους. Οι μέσες ηλικίε έχουν φύγει στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Και αυτό είναι πολύ θλιβερό. Ε, Έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δυο σας. Για αυτό που μας είπατε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτή τη χώρα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και μας είναι τόσο προσφυλής. Ευχαριστούμε πολύ. Bueno, vamos a ir rápidamente a las preguntas de los colegas. Eh... Λοιπόν, προχωρούμε. Sí, sí, sí. Señor Panceri, su pregunta. Κύριε Panceri, έχετε ερώτηση. La tua, la tua... Ερώτηση δεν έχεις, παιδάκι μου. Pregunta, questione, πώς το λες στα Ιταλικά, domanda. Sì, posso leggerla, sì, sì, Μπορώ να σας τη διαβάσω άμα θέλετε. Τα λέω εγώ. Well, it's a question on, on, on Tibet. I, I think that... Για το Θιβέτ. Εδώ είναι και ο εκπρόσωπος για να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Παντσέρη για το Θιβέτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώς υπάρχουν ε, πολλοί νέοι στο Θιβέτ οι οποίοι ε, εξακολουθούν να αυτοπιπολούνται. 141 κάτοικοι του Θιβέτ αυτοπιπολήθηκαν τον τελευταίο καιρό 114 από αυτούς μετά τη διαμαρτυρία τους έχασαν τη ζωή τους. Η ποινικοποίηση α, της α, διαδικασίας αυτής, η συνενοχή σε αυτή τη διαδικασία οδήγησε και σε θανατικές καταδίκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σε πολυμερές επίπεδο αλλά και διμερές επίπεδο την ανησυχία της. Η δήλωση της Γενικής Συνέλευσης θα έλεγα δείχνει τη στάση αυτή ζητάμε από τις κινέζικες αρχές να αντιμετωπίσει τις ε, βαθύτερες αιτίες της δυσφορίας των Θηβετιανών και ζητά να γίνονται σεβαστά τα πολιτιστικά και θρησκευτικά δικαιώματα. Θα πρέπει να υποστηριχθούν λοιπόν τα δικαιώματα των κατοίκων του Θιβέτ και να ελευθερωθούν όλοι όσοι συμμετέχουν σε παράνομες διαδηλώσεις. Έτσι θα μπορέσουν όλοι οι εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών και οι δημοσιογράφοι ελεύθερα να επισκέπτονται το Θιβέτ. Από την προσπάθεια του Δαλάη Λάμα το 10, τους εκπροσώπους του Δαλάη Λάμα δεν έχει υπάρξει επαφή από το 2010 επαναλαμβάνω και μετά να επιβεβαιώσω ότι τέτοια μηνύματα δόθηκαν στο υψηλότατο επίπεδο και στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου τον Μάιο και στη συνάντηση κορυφής τον Ιούνιο. Ο θάνατος στη φυλακή του Ντεν Σιν Ντεν Λεκ ε, δείχνει ακριβώς τι υποφέρουν οι κάτοικοι του Θιβέτ. Ο επόμενος διάλογος είναι τον μήνα Νοέμβριο με την Κίνα και θα θέσουμε εκ νέου τα θέματα αυτά. Sì, grazie. Capisco la risposta, ma mi pare... Κατανόησα την απάντησή σας, αλλά δεν βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε ένα ωραίο δώρο στον Δαλάη Λάμα για τα 80 του χρόνια. Θα πρέπει το θέμα αυτό να τεθεί με ε, πολύ αυστηρότητα προς τις κοινοζικές αρχές. Πέρα από το ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, φοβάμαι ότι όταν συνομιλούμε με τη συγκεκριμένη χώρα είμαστε σε θέση αδυναμίας, ενώ θα έπρεπε να εκφράσουμε από πλευράς Ευρώπης μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Πράγματι η φράση ελπίζουμε στον επόμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινέζικες αρχές είναι μια φράση την οποία θα έλεγα δεν έχει και πολύ περιεχόμενο. Όπως είπα, τα θέματα αυτά τίθενται στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο σε όλες τις διμερείς συναντήσεις μας με τους Κινέζους τέθηκαν και στα πλαίσια του στρατηγικού ε, διαλόγου και στα πλαίσια της συνάντησης κορυφής. Όχι με γενικούς όρους, αλλά με συγκεκριμένα ονόματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι κινέζικες αρχές, όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της συζήτησης, τόσο πιο ε, έμονοι είναι στις απαντήσεις τους, ότι έχουν τη δική τους άποψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρούν ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει βελτίωση στον τομέα αυτό, ακολουθούν το δικό τους δρόμο για την ανάπτυξη και έτσι κρίνουν την κατάσταση. Δεν αποφεύγουν τις ερωτήσεις, απαντούν στις ερωτήσεις στο υψηλότερο επίπεδο όπως είπα, αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν. δεν θεωρούν ότι πρέπει να απαντήσουν μόνο σε επίπεδο επί της αρχής, αλλά και με οικονομικά επιχειρήματα. Πάντως, επαναλαμβάνω, δίνουν πάντα την ίδια απάντηση μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόχ Μπίλε έχει ερώτηση για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, η ερώτησή μου έχει να κάνει με την ελευθερία της έκφρασης και το συνεταιρίζεστε από το 2011 ε, στα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εμείς εγκρίναμε ένα ψήφισμα το 2012 που το αναφέρουμε. Το 2013 στη συνέχεια 94 ακτιβιστές δικάστηκαν σε μια μαζική δίκη και 69 καταδικάστηκαν σε φυλάξη και κάθεξη μέχρι 15 χρόνια μόνο για μια ειρηνική διαδήλωση όπου εξέφρασαν τη γνώμη τους. Και ειδικοί ε, αναλυτές και εισηγητές στα Ηνωμένα Έθνη επιλήφθησαν και ε, τα αρμόδια όργανα ζητούν ε, άμεση και ανηφόρον ε, απελευθέρωση ε, των 94 που δικάστηκαν εκεί. Έχω έξι ερωτήσει εγώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της αναλαμβάνουν καμιά δράση μεταξύ αυτών παρατήρηση της δίκης για να αξιολογήσουν την μαζική δίκη και πώς διαβιβάστηκαν τα ευρήματά τους και τα πορίσματά τους και προς τις αρχές του τόπου και προς το κοινό γενικότερα και την κοινή γνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να αφαιθούν ελεύθεροι 69 καταδικασμένοι κρατούμενοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει να ζητήσει δημόσια να αφαιθούν ελεύθερα και, ελεύθεροι και ανεφόρων ως ε, κρατούμενοι συνείδησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει να επισκεφθούν κανέναν από τους 69 κρατουμένους στη φυλακή. Και αν ναι, εγκρίθηκαν αυτές οι επισκέψεις και τι διαπίστωσαν. Προτίθεστε να προβείτε σε καμιά περαιτέρω δράση ή επίσκεψη. Και μια πιο γενικότερη ερώτηση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 14ος ε, μεγαλύτερος διεθνής εταίρος. Εμπορικός εταίρος με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τι κάνει για να αξιοποιήσει αυτή τη θέση της γενικά στη χώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σλόβεκ θα απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορώ να απαντήσω και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να πω ότι μετά από την υιοθέτηση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου το 12 τα Εμμυράτα αντέδρασαν οργήλως βασιζόμενοι στην προτινόμενη λύση και στο ψήφισμα αυτό και στις εξελίξεις στη Γενέβη και την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ανεπίσημη ομάδα εργασίας. Είναι το φόρουμ στο οποίο έχουν συζητηθεί τα θέματα αυτά τελευταία Πιο συγκεκριμένα τώρα έρχομαι στις ερωτήσεις σας. Σχετικά με την μαζική δίκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποστολή στο Αμπουντάμπι ζήτησε τον τίτλο του παρατηρητή, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό. Το θέμα των 69 φυλακισμένων είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται συστηματικά από όλες τις πλευρές και στην παρούσα φάση δεν ε, ζητάμε δημόσια την απελευθέρωσή τους, αλλά προσπαθούμε με σιωπηλό δημοκρατικό τρόπο να την πετύχουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πρακτική να επισκέπτεται ε, τους φυλακισμένους. Στα πλαίσια της τελευταίας ανεπίσης ομάδας εργασίας το ζητήσαμε, μας έδωσαν την δυνατότητα αυτοί επέλεξαν σε ποια μονάδα κράτησης θα μας οδηγούσαν, δεν μας πήγαν στο Αλαραζάν όπου κρατούνται οι 69. Και γι' αυτό εμείς πιθανώς στο μέλλον θα ζητήσουμε μια άλλη συνάντηση ε, στα Εμμυράτα για να επισκεφθούμε και κάποια άλλη τέτοια μονάδα. Και ελπίζω σε αυτή την περίπτωση να μας δοθεί άδεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γνωρίζει αδίποτε επίσκεψη ε, κρατών μελών στη φυλακή. Στο κέντρο κράτησης δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες και η αδίποτε δράση ε, θα αναλυφθεί έτσι ώστε με τις αρχές των Εμμυράτων σε διπλωματικό επίπεδο ε, να προωθούμε την ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, και να ζητήσουμε για μια ακόμη φορά από τους εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών να μπορέσουν να επισκεφθούν τη χώρα και να συνεργαστούν οι αρχές των Εμμυράτων μαζί τους. Τελευταία ερώτηση σχετικά με την οικονομική επιρροή. Εμείς έχουμε μια αντιπροσωπεία στο Αμπουντάμπι στο τέλος του 2013. Τώρα η αντιπροσωπεία αυτή προσπαθεί να συντονίσει και να ενισχύσει τις θέσεις των κρατών μελών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Να αναφέρω επίσης ότι η εξωτερική υπηρεσία έχει κάποια διπλωματικά μέσα στη διάθεσή της, αλλά να μην ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ περισσότερη επιρροή και θα πρέπει και αυτά να τους ζητηθεί να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους προς τις ε, αρχές των Εμμυράτων ιδιαίτερα ε, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η διαδικασία εξαίρεσης από την υποχρέωση έκδοσης θεωρήσεων ήταν κάτι το πάρα πολύ θετικό για τα Ηνωμένα Εμμυράτα. Ευχαριστώ. Δεν είναι μαζί μας ο κύριος Χάινκελ, αλλά ο κύριος Δεμέρς Μέκερ μπορεί να θέσει την ερώτησή του. Για τους Ροχίνγκα, να η ερώτηση του Χάνκελ είναι τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα των Ροχίνγκα. Νομίζω ότι θα απαντήσει η κυρία Νέμεθ. Έχετε το λόγο. έχετε το λόγο. Okay, yes. Thank you very much uh, for the, uh, for the European Parliament. ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ και ιδιαίτερα για τους Ροχίνγκα. Το θέμα είναι από τα κυριότερα για την Ένωση στον διάλογό της με τη Μιανμάρ. Στις 22 Ιουνίου το Συμβούλιο Εξωτερικών στα συμπεράσματά του για τις ε, επικείμενες εκλογές στη Μιαμάρ ή η Βυρμανία αναφέρει ότι η αναφερει οτι ζητάει διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές τις οποίες να μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι κάτοικοι της Μιανμάρ ακόμη και οι μειονότητες για να ασκήσουν έτσι το εκλογικό τους δικαίωμα ελεύθερα. Στις τα ίδια συμπεράσματα του Συμβουλίου τονίζεται ότι η λύση για το θέμα της ηθαγένειας των Ροχίνγκα, η λύση του προβλήματος θα συνέβαλε στη λύση της ε, μεταναστευτικής κρίσης στην περιοχή και θα έσωζε ζωές και δουλεμπόριο. Κατά την επίσκεψη στη Μιανμάρ στις 14 με 18 Ιουνίου ο ειδικό εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Εσταύρος Λαμπρινίδης επίσης έθεσε το θέμα των Ροχίνγκα με τους ε, πολιτικούς που συνάντησε εκεί, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Πληθυσμού και τον κύριο Υπουργό του κράτου Ιδίου Ρακάν. Με όλους αυτούς ζητήθηκε να βρεθεί μια λύση για τον πληθυσμό που ζει σε εκείνα τα μέρη επί πολλούς αιώνες και ζήτησε συνεργασία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο ΡΑΚΑΝ για να τονιστεί η σημασία της εξέβρεσης στα δικαιώματα των μειονοτήτων καθώς και των Ροχίνγκα συζητήθηκαν και στο δεύτερο διάλογο Ένωσης Μιανμάρ 18 Ιουνίου που έγινε στον Έπιτον. Εκτός αυτού, η Ένωση συνεχίζει να καταθέτει ψηφίσματα για την κατάσταση των δικαιωμάτων στη Μιανμάρ και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο κρατήδιο του Ρακάν η κατάσταση συζητιέται και σε πολλά ψηφίσματα παρά το δύσκολο περιβάλλον εργασίας των οργανώσεων του ΙΕ, οι δικαιοδοσίες τους έχουν αυξηθεί και σήμερα η Ένωση, η Ένωση είναι από τους κυριότερους παράγοντες που δρούν στο κρατήδιο του Ρακάν, τονίζοντας ιδιαίτερα θέματα παιδείας, υγειονομικά, συμφιλίωσης και καταπολέμησης της άνησης μεταχείρισης. Η βοήθεια που δίνουμε εκεί ξεπερνάει τα 35 εκατομμύρια κυρίως ανθρωπιστικής βοήθειας. Εκτός από τη βοήθεια που δίνουμε στους Ροχίνγκα, η Ένωση επίσης χορηγεί ανθρωπιστική βοήθεια για πρόσφυγες Ροχίνγκα στην Μπαγκλαντές και επίσης βρίσκεται σε στενές επαφές με τις αρχές στην Ταϊλάνδη με την οποία έχει ενδυναμωθεί ο διάλογος για την κατάσταση των Ροχίνγκα. Οι αρχές της Ταϊλάνδης έχουν πάρει ορισμένα μέτρα όπως καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου και ανακάλυψη μαζικών τάφων. Η κυρία Μογκερίνη επίσης είναι γνώστης του θέματος των μαζικών τάφων και των Ροχίνγκα και έγραψε μία επιστολή στον Υπουργό Ιστορικών Τανασάκ 26 Μαΐου. Η Κομισιόν πρόσφατα έχει χορηγήσει νέα πόρους 300.000 ευρώ για τη στήριξη των Boat People Rohingya και στην Ινδονησία και στη Μαλαισία. Εκτός αυτού, η Πάτη Μογκερίνη έθεσε και το θέμα της μεταναστευτικής κρίσης Ευρώπης και Νοτιοανατολικής Ασίας στις 29 και 30 Μαΐου και τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η διάσωση ζωών και η λύση του προβλήματος στη ρίζα του. Επίσης τόνισε την ανάγκη να καταπολεμηθεί το τουλεμπόριο στις χώρες διαμετακόμισης και προέλευσης. Η συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την εξέβρεση λύσης είναι επίσης ουσιαστική χωρίς να ξεχνάμε το θέμα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και του εμπορίου ανθρωπίνων όντων καθώς και του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Τελεία. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μάρκ, έχεις να προσθέσεις τίποτα. Ναι. Όχι πάρα πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ε, απάντηση. Τα σημαντικότερα τα σημείωσα mm -hmm. και θα τα πω και στον κύριο Χένκελ, θα τα διαβιβάσω. Ο οποίος ο κύριος Χένκελ είναι ο συντάξης ερώτησης. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε τη τελευταία ερώτηση του κυρίου Στρεβίτσιους. It is very clear, Είναι σαφέστατη ερώτηση, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω. Μάλιστα, μπορείτε να απαντήσετε κύριο Μπράιαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει το θέμα των βασανιστήριων στις ε, συναντήσεις που έχει για το διάλογο με τις χώρες Κεντρικής Ασίας. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αφιερώσει ειδική ε, ατζέντα σε όλες ε, τις χώρες και στο διάλογο που είχαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το Τουρκμενιστάν και το Τατζικιστάν τον περασμένο μήνα με την Δημοκρατία της Κυργυζίας το Μάιο και το Καζακστάν και το Ουσπεκιστάν τον περασμένο Νοέμβριο. Βεβαίως ε, θέτουμε πάντα αυτό το θέμα προσώπων που έχουν φυλακιστεί γιατί είχαν πολιτική ειρηνική δράση ε, και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές κλπ. Ε, κάνουμε και συστάσεις στις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής για την πρόληψη των βασανιστήριων και βεβαίως διαφέρουν οι συστάσεις ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα σε ορισμένε περιπτώσει έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την πρόληψη των βασανιστήριων οι κυβερνήσει και τι υποστηρίζουμε και τι ενθαρρύνουμε, ενώ σε κάποιε άλλε ε, η πρόοδο ήταν πολύ βραδύτερη. Δεν υπάρχει ένα μέτρο που να συστήνουμε σε όλα τα κράτη για την πρόληψη των βασανιστήριων. Ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις εταίρους μας να προβούν σε μεταρρυθμίσεις και πολιτικής και νομοθεσίας για να έχουμε ουσιαστική μείωση και εξάλληψη των βασανιστήριων. Ορισμένα από τα συγκεκριμένα βήματα που προτείνουμε είναι νομοθετική μεταρρύθμιση έτσι ώστε να είναι ιδιώνυμο ε, ε, το βασανιστήριο και ε, να μην χρησιμοποιούνται στοιχεία που έχουν αποσπαστεί μετά από βασανιστήρια στα δικαστήρια κατά τη διάρκεια της δίκης ε, ανεξάρτητοι μηχανισμοί με, με σωστή στελέχωση και ε, χρηματοδότηση, εκπαίδευση για την πρόληψη των βασανιστήριων για τις διοκτικές αρχές και τις δικαστικές αρχές νέα μέτρα για την καταχώρηση κρατουμένων σε αστυνομικά τμήματα, πρόσβαση σε δικηγόρους από τα πιο πρώιμα στάδια της ε, κράτησης, ε, συστήματα παρακολούθησης σε κελιά και σε ανακριτικά γραφεία, ε, συνδρομή ιατρική και νομική σε θύματα βασανιστήριων. Επίσης, για την ατιμορρησία κάνουμε συστάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι καταγγελίες βασανιστήριων να ε, ε, παρακολουθούνται, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να δίνεται συνέχεια και σε ό,τι αφορά τις διοκτικές αρχές θα πρέπει οι να σέβονται, ή υπάλληλοι ε, να σέβονται και να υπακούν στους νόμους. Είναι μεικτή πάντως η εικόνα στην περιοχή, δεν είναι ενιαία σε όλες τις χώρες και πραγματικά πρέπει να πούμε ότι δεν δίνεται πραγματική συνέχεια συχνά στις καταγγελίες. Ε, σε όλη την περιοχή χρειάζεται προσπάθεια. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει ένα τριετές πρόγραμμα με το Ίδρυμα του Ελσίνκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 1,1 εκατομμύριο ευρώ είναι ο προπολογισμό για την πρόληψη βασανιστήριου στο Τατζικιστάν και στο Καζακστάν το 2013. Άλλο τριετές για τα παιδιά και τις φυλακές αντιλίκων από ε, μια διεθνή οργάνωση για την ποινική μεταρρύθμιση ε, που έχει να κάνει με το Κασαχστάν, ε, το Τουρκμενιστάν και το Τατζικιστάν 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Με την Κυρχησία είναι το πέμπτο σεμινάριο τον Οκτώβριο, ειδικά για την πρόληψη των βασανιστήριων με 70 εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών ε, από νομικά επαγγέλματα, το διαμεσολαβητή, το συνήγορο του πολίτη, το ανώτατο δικαστήριο, Υπουργείο Εστερικών και άλλους κρατικούς φορείς. Επίσης, χρηματοδοτούμε διάφορα έργα στην Δημοκρατία της Κυργυσίας ε, και σε συνεργασία με ε, εθνικές αρχές χρηματοδοτούμε και προωθούμε αυτά τα θέματα. Αυτά είναι λίγα παραδείγματα μόνο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή και ε, να πιέζουμε για περαιτέρω πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αουστρεδίτσιος Σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτές τις πληροφορίες. Το θέμα παραμένει στην ημερήσια διάταξη των ε, ανωτά των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν επισκέπτονται την περιοχή. Θα ήθελα τις πληροφορίες αυτές να τις αποστείλετε και στην αντιπροσωπεία με τις δημοκρατίες των χωρών της Κεντρικής Ασίας για να το συζητήσουν και αυτές είναι πληροφορίες ε, τις οποίες μας είπατε χρήσιμες και ακόμα περισσότερες μπορείτε να μεταφέρετε διότι η κατάσταση ως έχει δεν είναι διόλου ικανοποιητική και είναι σαφές ότι υπάρχουν βασανισμοί και μορφές κράτησης που προσωμιάζουν στο βασανισμό για τους πολιτικούς κρατημένους ίσως και για άλλους κρατημένους, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για μας. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος στην επιμελητία. Καλό καλοκαίρι και προς τους διερμηνείς. Ευχαριστώ. 22 Σεπτεμβρίου η επόμενη συνεδρίαση.